Ja, guten Tag. Ja. good afternoon. Καλησπέρα σας λέει η Πρόεδρος. Αν θέλετε να αρχίσουμε τη συνεδρίαση στα γερμανικά. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Δεν έχει καταθέσει κάποιος δύο οπότε εγκρίνεται ω έχει. Στο σημείο 2 βλέπετε τις γλώσσες οποίες υπάρχει διερμηνία και όσοι ήθιστε μεταδίδετε στο διαδίκτυο. Ε, παρακαλώ να προετοιμάσετε τις ε, κάρτες ε, για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και ε, βρείτε τις αν δεν τις έχετε φέρει ακόμη, σημείο 3. Ε, να εγκρίνουμε τα πρακτικά από τις προηγούμενες ε, συνεδριάσεις από Ιανουάριο και Φεβρουάριο, έτσι. Και ό συνήθω, αν δεν προβάλλεται ενστάσεις μέχρι το πέρας συνεδρίας, εγκρίνονται. Ε, σημείο 4 και αρχίζουμε με Αρχίζουμε, τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται, τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση. Ε, άρχεται ψηφοφορία. Το Πέρας. Είναι ακόμη ανοιχτή η ψηφοφορία. Δεν έχουμε ψήφους κατά. Με 20 ψήφους ε, εγκρίνεται. Για πάμε τώρα στο ψήφισμα. Για την απαλλαγή. Όχι, όχι. Για την απαλλαγή ήταν το προηγούμενο. Πάμε. Για, ε, τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είμαστε στο ψήφισμα κοντ τώρα. Αυτό σε Αυτό και πάμε τώρα στο ψήφισμα, σημείο 3, ε, τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Μπορούμε να, να επαληθεύσουμε για τροπολογία 6 παρακαλώ. Δύο κάρτες βλέπω δεν έχουν ψηφίσει.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 Επαλήθευση παρακαλώ για τη 43. 43 επαλήθευση. Πέρας, εγκρίθηκε. 44 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επαλήφθηση για την 50 σας παρακαλώ πολύ 50 Έχουμε ακόμη πέντε κάρτες που δεν έχετε ψηφίσει. Α, τώρα εντάξει, πέρας. Α, απορρίπτεται. Ναι. Συμβαστική 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε. Τις συναρμόδιες επιτροπές, ΔΒ1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΒ2 υπέρ Καλύπτεται DV3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται DV4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται DV5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται DV6 υπέρ, κατά απο... Ξανά, για την DV6 υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Επαλήθευση DV6. Πέρασε. Απορρίπτεται δε 7 υπέρ κατά αποχές. Τι είναι αυτό τώρα ΔΕΒ7 υπέρ απόχέ. αποχές. δβ ΔΕΒ8 υπέρ κατά. ΔΕΒ8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ε, τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται. Ονομαστική ψηφοφορία. Εγκρίθηκε με 17 ψηφού ε, Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ε, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία. Στο και αν δεν κατάλαβα πολύ καλά, γιατί οι σοσιαλιστές συνάδελφοι συμμετείχαν εδώ. Λοιπόν, ε, τώρα δίνω το λόγο στον εισηγητή. Θα είμαι πολύ σύντομος θα ήθελα να ζητήσω από τους συνεδέλφους να ακολουθήσουν τις συστάσεις μου όσον αφορά τη ψηφοφορία, γιατί πιστεύω ότι είναι όλες πολύ λογικές. Μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή την επιθυμία. Αυτή την επιθυμία έχουν πολλοί, άλλωστε. Συμφωνώ με τον κύριο Βον, αλλά θέλω να σας πω ότι όσον αφορά τις γλωσσικές εκδοχές ισπανική συγκεκριμένα, υπάρχει λάθος μετάφραση για αυτούς τους βοηθούς συνεργάτες ε, που είναι πάντοτε διαπιστευμένοι και στο 108 υπάρχει ε, ένα λάθος γιατί λέει για τα εσωτερικά μέλη, εσωτερικούς βουλευτές ε, και εννοεί κάποιους που έχουν τύχει υποτροφίας να προσέξουμε να γίνει διόρθωση χτένισμα της μετάφρασης της, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνίες και να λιωθεί μετά τελικά η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ για την επισήμανση και τώρα θα έρθουμε στην απόφαση για την απαλλαγή. Η τροπολογία υπαριθμών 1, 1 και 2 μάλλον από κοινού, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, στην απαλλαγή, για την απαλλαγή ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας της ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 22 κατά, χορηγείται η απαλλαγή. Τώρα θα έρθουμε στο ψήφισμα. Ε, 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές. Μπορούμε να το ελέγξουμε την 4 παρακαλώ. Πέρας του ελέγχου εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 είναι συμβατή, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, καταπίπτει. 16 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 17 με, την, με προφορική τροπολογία δεν υπάρχουν ενστάσεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ α, σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ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 πέρας της επαλήθευσης ε, απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, θα είναι νομίζω η ίδια, το ίδιο ποσοστό. Το δεύτερο τμήμα, το επαληθεύσουμε. Τροπολογία 25. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 26 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ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 αποχές επαλήθευση για την τροπολογία υπαριθμών 34. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ για τη 39, 39 ε, συγγνώμη, ε, σε κατά τμήματα, σε δύο τμήματα. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε τώρα split ε, vote. Υπάρχουν κάποιες προθεσμίες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 132 υπέρ, α όχι <laughs> καταπίπτει, 40 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται, 41 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Συμβασμός παρθούν 1 υπέρ, κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση 1, συμβαστική 1. Πέρας της ηλεκτρονικής επαλήθευσης εγκρίνεται 42 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ 49 και 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Ωραία. Θα γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση για την ε, συμβαστική 50. Πέρας της επαλήθευσης εγκρίνεται. Τρία συμβαστική ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 54. Με προφορική τροπολογία δεν υπάρχουν στάσεις υπέρ, κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την 54 με προφορική τροπολογία. Πέρας της ε, επαλήθευσης απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά απορρίπτεται. Για την 55 ηλεκτρονική επαλήθευση. Ωραία. Τέλος της εγκρίνεται. 56 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 για την 56 επαλήθευση. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ξεκάθαρη η πλειοψηφία. Τέλος πάντων, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Πρώτο τμήμα, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει λέει η πρόεδρος. 60 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την υπαριθμόν 60. Τέλος της ηλεκτρονικής επαλήθευσης εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται 62 υπέρ, κατά, απορρίπτεται 63 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται 64 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται 65 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται 66 υπέρ, κατά αποχές, θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση για την 66, δεν ήταν ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. τέλος της, ε, του ελέγχου ε, εγκρίνεται. Ε, η 64 καταπίπτει, 68 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 69 καταπίπτει, ναι, καταπίπτει 69, έχουμε την 70 υπέρ, κατά αποχές. Απορρίπτεται 71 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 72 επέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 κατά πίπτη 73 επέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 επέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 Α, όχι, 76. 76, 76 την ψηφίσαμε, 77. Υπέρ κατά αποχές την 77 να επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφορία ωραία απορρίπτεται συγγνώμη ε, 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 83 εγώ πιστεύω ότι απορρίπτεται αλλά εν πάση περιπτώσει απορρίπτεται ευχαριστώ 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ όχι, καταπίπτει λέει η πρόεδρος, 86 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ, κατά αποχές επαλήθευση για την 87. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεται. 88 υπέρ. Ναι, είναι συμβατή με την 86 και την 87. 88 υπέρ, κατά, αποχές, υπέρ. Πάλι υπέρ, κατά, αποχές. Ωραία, ηλεκτρονική επαλήθευση την 88. εγκρίνεται 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές 92 επαλήθευση εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 96 Εγκρίνεται 97 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ,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 Δέκατο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δέκατο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται κατά την άποψή μου. Επαλήθευση για την 103. Το beendet. Πέρασης ε, του ελέγχου εγκρίνεται 104 κατά 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 σε 8 τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Έκτο τμήμα υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Έβδομο τμήμα υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Όγδο τμήμα υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Και τώρα 109 με προφορική τροπολογία. υπάρχει μια ένσταση κατά της προφορικής τροπολογίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το πρωτότυπο κείμενο λέει η πρόεδρος μάλιστα ακριβώς ε, απορρίπτεται το αρχικό κείμενο το αρχικό κείμενο 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 118, α, 120, συγγνώμη, υπέρ, κατά αποχές 120, έλεγχος. Τέλος του ελέγχου εγκρίνεται 117 υπέρ. Όχι, καταπίπτει. 121 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 125 και όχι πίπτη, 129 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται 130 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 131 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 131 πρώτο τμήμα. Απορρίπτεται. 131 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται θέλετε να γίνει επαλήθευση για την 134 παρακαλώ εγκρίνεται όχι απορρίπτεται απορρίπτεται 135 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για το πρώτο τμήμα της ε, υπαριθμών 136 εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, Σεβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ, α όχι καταπίπτει, 140 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 145 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ, 150 συγγνώμη, υπέρ κατά εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά 158 50. Der Check ist beendet. Das ist angenommen. Α, εγκρίνεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση για την 163 υπέρ. Ε, όχι, συγγνώμη, <laughs> ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας της ε, επαλήθευσης απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα ελέγξουμε τη συμβαστική παριθμόν 8 εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση 179. Πέρασε επαλήθευση. Εγκρίνεται. Συγγνώμη, δεν το είδα, λέει η πρόεδρος. 180 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 181 υπέρ Κατά αποχές απορρίπτεται 182 υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση 182. Πέρα της επαλήθευση, εγκρίνεται 183 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 184 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 185 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 186 Καταπίπτει. 187 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 193 καταπίπτει. 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 201 έχει αποσυρθεί 202 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 204 υπέρ. Κατά επαλήθευση για τη 204. Πέρασε επαλήθευσης. Εγκρίνεται 205 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 206 υπέρ. Κατά αποχές Μπορεί να γίνει επαλήθευση για την υπαριθμό 206, παρακαλώ. Πέρασε τη εφορία. Εγκρίνεται. 207 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται 208 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται 209 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 210 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 213 υπέρ κατά αποχές παρακαλώ να γίνει επαλήθευση για τη 213 απορρίπτεται με ισοψηφία και τώρα έχουμε στη τελική ψηφοφορία, ονομαστικά, με ονομαστική κλίση για το ψήφισμα στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία 19 προς 3. Θερμά συγχαρητήρια προς τον εισηγητή. Damit sind wir am Ende der Abstimmungen. Die... Ολοκληρώσαμε τις ε, ψηφοφορίες ε, του εξωτερικού οργανισμού. Αύριο θα τους ψηφίσουμε. Please. <laughs> for the coordinators, for the coordinators we start. When we are ready with the meeting, we start immediately. Για τους συντονιστές θα αρχίσουμε με το που είστε έτοιμοι γιατί έχουμε πάρα πολύ βάρια ημερήσια διάταξη. Ja, damit wir kommen zum Sonderbericht 5 2018. Ε, περνάμε τώρα στην ειδική έκθεση 5 του 2018 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη της ε, ε, υπαίθρου. Η εισηγήτρια η κυρία Κάντεμπαχ και η παρουσίαση από τον κύριο Γέρεπ. Γεια σας κύριε Γέρεπ. Παρακαλώ όμως να ησυχάσετε για να μπορέσουμε να ακούσουμε την παρουσίαση. Wir haben, Kurzvorstellungen. παρουσίαση, κύριε Γέρε, παρακαλώ. Thank you, Madam Chair. Honorable members of the committee. Πρόεδρε, βουλευτέ, ευχαριστούμε μας την ευκαιρία να ε, τα συμπεράσματα της Επιτροπής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ε, συνέργειας κλπ. Πρόκειται για μια ενέργεια από πηγές ενεργειακές, παραδοσιακές, απορρικτά κάψουμε δηλαδή, αλλά επίσης έχουμε να κάνουμε ακόμα πολλές προσπάθειες αν θέλουμε αυτούς τους στόχους του 20% από ανανεώσιμες μέχρι το 2020 να το πετύχουμε με το 27% του 2030. Και όλα αυτά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τη Συμφωνία των Παρισίων για την αλλαγή του κλίματος. Και επίσης έχουμε κάποια άλλα προγράμματα, ούτως ώστε να δοθούν κίνητρα για την παραγωγή και ε, πηγή πόρων ε, αφορά και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης. Οπότε εξετάσαμε τη σχέση μεταξύ ανανεώσιμης ενέργειας και αγροτικής ανάπτυξης, να ανανεώσουμε ενέργεια συνολικά και πώς αυτά ενσωματώσαν κάποιες πτυχές αγροτικής ανάπτυξης και καταλήξαμε ότι υπάρχουν συνέργειες για την ε, αγροτική ανάπτυξη, για την, ε, την ανάπτυξη ανανεώσιμης ε, ενέργειας, αλλά λόγω συνέργειες έχουν παραμείνει αναξιοποιητές και διάφορες αυτές αφορούσαν τις πολιτικές για να βελτιωθεί η κατάσταση. Όμως ούτε το σημερινό πλαίσιο ούτε το προτινόμενο μας έδωσαν μια αρκετή βάση ούτω ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε από τους κινδύνους ή να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να συμβάλλει για την ανάπτυξη ε, των αγροτικών περιοχών. Όμως, ακόμη δεν έχει δοθεί προτεραιότητα στα έργα που θα έπρεπε. Ούτε η Επιτροπή έχει επαρκή στοιχεία για τις δαπάνες του Ταμείου Αγροτικής ανάπτυξη για αυτή την ε, ανανεώσιμη ενέργεια. Οπότε, τα περισσότερα κράτη-μέλη τα οποία επισκεφθήκαμε δεν έδωσαν προτεραιότητα σε αυτά τα προγράμματα. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2017, δηλαδή, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολιετού δημοσιογραφικού πλαισίου, είχαμε μόνο το 5% της έκτασης που λοιπόν να αξιοποιηθεί. Και έτσι φτάσαμε στην περίοδο 2017-2013. Και δεν υπήρχαν τα στοιχεία για το πόσο όλα αυτά καλύφθηκαν στις σχετικές δαπάνες και επίσης υπήρχαν λίγες πληροφορίες για το τι έγιναν οι πόροι που διατέθηκαν παρά τις πρόοδους. Το 2014-2020 ακόμα έχουμε αδυναμίες στο, στην περίοδο προγραμματισμού και επίσης ως αυτό το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής των βασικών δικτών. Στο δείγμα που ελέγξαμε είδαμε τις επενδύσεις για παροχή σε τρίτους ανανόσιμων πηγών και επενδύσεις για παραγωγή ενέργειας για ίδια κατανάλωση. Θεωρήσαμε τα περισσότερα έργα ήταν πετυχημένα γιατί υπήρχε οικονομικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος για την ανάπτυξη. Όμως, αδυναμίες στην επιλογή επίσης κάνουν στο αποτελέσμα των έργων που έδωσαν όφελο στους κύριους των έργων αλλά όχι στις ε, αγροτικές περιοχές και επί τη βάση αυτό να διαπιστώσεων έχουμε γράμμα τις εξής συστάσεις. Η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη Πρέπει να λέει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών, ιδίω όταν καταρτίζονται τα εθνικά σχέδια και με τους συνομοθέτες να φτιάξει ένα πλαίσιο πολιτικής για βιοενέργεια. Περισσότερες διασφαλίσεις για τη μη βιώσιμη χρήση των πόρων βιομάζας. Πρέπει να προσδιορίσουμε το σκοπό και τον ρόλο της παρεχόμενης στήριξης για αυτές τις επενδύσεις. Και θα πρέπει τα κρατημέλη να παράσχουν πληροφορίες για τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων. Και επίσης σε σχέση με τις ενισχυμένες αιτήσεις εκθέσεις υλοποίησης. Να εφαρμοστούν κατάλληλες διαδικασίες επιλογής για να υποστηριχτούν μόνο βιώσιμα για την ανανεώσιμη ενέργεια που να ωφελούν την αγροτική ανάπτυξη. Ευχαριστούμε και θα απαντήσουμε τις ερωτήσεις, αν τυχόν υπάρχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σημαντική η έκθεση. Ε, βλέπουμε τι θα έπρεπε να γίνεται στην Ήπεθρο. Η κυρία Λωρίς Χόφων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την ε, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας θα πάρει το λόγο. Παρακαλώ κυρία μου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε μα δίνετε να ανταλλάξουμε απόψει για αυτή την ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για τι Ανανεώσιμε Πηγέ Ενέργεια για την Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη. Καλωσορίζουμε αυτή την ειδική έκθεση. Και επί ουσία έχουμε εγκρίνει τι ε, συστάσει του Ελεκτικού Συνεδρίου παρότι υπάρχουν κάποια σημεία, δεν μπορούμε να προδικάσουμε ακριβώ. Ε, με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο μετά το 2020 θα ε, επεξεργαστεί αυτά τα στοιχεία μέσα στις μελλοντικέ ε, νομοθετικές προτάσεις της. Για κάποια από τα ζητήματα που ήγηρε το ελεκτικό συνέδριο, θέλω και εγώ να κάνω σχόλια για την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, παρέχεται σημαντικό περιθώριο ελιγμών στα κράτη-μέλη για την επίτευξη του στόχου, μεταξύ των οποίων και ε, της χρήσης και πρόθεσης της, ε, της χρήσης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στην Ήπεθρο. Έχουμε το βιώσιμο πλαίσιο για τη βιοενέργεια που λειτουργήσε αποτελεσματικό για να αποφύγουμε τον έμεσο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Πρόσθετα μέτρα ελέγχθησαν το 2015 Επίσης, για να αντιμετωπιστεί ο Ιωνί ε, έμεσος ε, η πρόταση για την αναθεώρηση της ε, ισχύουσας οδηγίας ενισχύει σημαντικά αυτό το πλήσιο και παρέχει επιπρόσθετα ηχέγγυα για, την, για τον μη βιώσιμο εφοδιασμό δασικής βιομάζας για τα κριτήρια της ε, βιωσιμότητας βιοενέργειας δεν θα πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα διότι είναι ε, ε, συμπληρωματικά σε σχέση με άλλα, άλλες νομοθετικές πράξεις παραδείγματος χάρη αναθεωρημένη πρόταση για την χρήση της γης και τη δασοκομεία LUCF. Για τη χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας αναγνωρίζουμε φυσικά Μάλλον καλωσορίζουμε τότε το ελεγκτικό συνέδριο αναγνωρίζει πως έχει δυναμικό η ανανόσιμη ενέργεια για να συμβάλλει στην ανάπτυξη της υπαίθρου κυρίως με την συμμετοχή των τοπικών εταίρων και διαθέσιμη χρηματοδότηση για την αγροτική ανάπτυξη έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για τη χρήση ανανόσιμων μορφών ενέργειας. Στα πλαίσια της ανακοίνωσης για το μέλλον της γεωργίας και της διατροφικής πολιτικής Έχουμε δει την πρόθεση να ε, ενισχύσουμε τις δράσεις ε, στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος ε, με την μείωση της βιομάσας για όλες τις χρήσεις, ακόμη και για την παραγωγή της βιοενέργειας, για τη μελλοντική πολιτική ανάπτυξη πέθρου θα πρέπει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των εδαφών, όμως θα πρέπει να τονίζουμε πως η περιοχές των κρατών μελών είναι στην καλύτερη δυνατή θέση για να ε, προτείνουν και να αποφασίσουν πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο ως προς ε, τις επενδύσεις. θα υποστηρίξουμε τις αποφάσεις των κρατών μελών. Παραδείγματος χάρη με τη διάδοση των καλών πρακτικών βάση της ε, πολιτικής για την ανάπτυξη υπαίθρου στην ιστοσελίδα του δικτύου για την ανάπτυξη υπαίθρου. Εκεί δίνουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Πώς ε, δηλαδή ε, δυνατότητες και πώς ε, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό της χρήσης των ανανεώσιμων ενέργειας, αλλά και συνεργαζόμαστε με ομάδες κρατών μελών για την πρωτοβουλία ε, για, την, ε, για τις ε, καινοτόμες δράσεις έχουμε συστήσει μία ομάδα για την, τα διαθέσιμα ταμεία για τη χρηματοδότηση των δράσεων τον Νοέμβρη στάθηκε αυτή η ομάδα. Επίσης προτείνει το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η προσθέμενη αξία των προγραμμάτων των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η επιλογή των προγραμμάτων συνιστά αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία προσδιορίζουν ως εκ τούτου και τα κριτήρια επιλογής των προγραμμάτων. Τούτου λεχθέντος συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και για τον προσδιορισμό των κριτηρίων και για να συνδέσουμε τα κριτήρια με συγκεκριμένους στόχους και ακριβώς έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ήρθε και η συγγήτρια στο μεταξύ, η κυρία Κάντεμπαχ. Άμα θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ναι, ε, λυπάμαι που μιλάω μετά την παρουσίαση της έκθεσης. Ε, είναι ανάκατη συζήτηση, αλλά τέλος πάντων ε, είναι, είναι πολύ δύσκολο να είναι ε, εύστοχα τα σχόλιά μου λόγω χρονικού περιορισμού, επειδή έφτασα αγροπορημένη. Ευχαριστούμε λοιπόν παρά όλα αυτά ε, για την αποφασιστική σημασία σε έκθεση για το μέλλον της γεωργικής πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020 και είμαστε ευγνώμονες και ε, επιμένουμε ότι πρέπει να έχουμε επαληθεύσιμα ε, κριτήρια για να διαμορφώσουμε τη μελλοντική γεωργική πολιτική και ε, υπάρχουν και θέματα που φυσικά εκφεύγουν τις αρμοδιότητες μας Όταν μιλάμε για τα ισοδύναμα του διοξιδίου του άνθρακα, παραδείγματο χάρη για την ανακοίνωση ε, τη Επιτροπή, ε, βλέπουμε ότι ε, όποια μέτρα λαμβάνονται έχουν, είναι αλληλοσυμπληρούμενα, έχουν άμεσα, άμεσες επί των υπολείπων και όλα επηρεάζουν την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη... Πρόσφατα συμφωνήσαμε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά τα ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου είναι ένα μεμονωμένο θέμα και μεμονωμένο και η προστασία του περιβάλλοντος ε, ή τα μέτρα για την αντιμετώπιση των αλλαγών του κλίματος. Όλα σφαιρικά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, να ε, ομαδοποιήσουμε τα μέτρα. Και το βλέπουμε μέσα στην έκδοση ότι κάποια μέτρα που λαμβάνονται σε ένα πυλώνα, σε ένα σιλό και έχουν θετικό, ε, θετική επίπτωση όταν τα εξετάζουμε, γενικότερα βλέπουμε ότι δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ε, Παραδείγματο χάρη, όταν κάτι είναι θετικό, ε, μια προμοδότηση για την γεωργική χρήση της γης, ε, όταν εξετάζεται σφαιρικά σε σχέση με την ανάπτυξη της υπαίθρου και της ευρύτερης περιοχής, διαπιστώνουμε ότι το μέτρο δεν είναι τόσο θετικό. Οπότε, ε, ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν και όχι να ε, εξασφαλίσουμε μόνο τις πηγές εισοδήματος των μεμονωμένων δικαιούχων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε ένα έγγραφο εργασίας και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε και στο μέλλον να ζητήσουμε διεξοδικότερα αυτή την έκθεση, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να συμπληρώσουμε με τις παρατηρήσεις μας ε, φυσικά είναι ιδιαίτερα σημαντική η έκθεση διότι το θέμα της ανάπτυξης και το θέμα ε, της ενέργεια ενέργειας ε, είναι θέματα που συνδέονται άμετα με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό το έγγραφο εργασίας άρα είναι εξαιρετική ευκαιρία για να οριοθετήσουμε, να προσδιορίσουμε και εμείς τη θέση μας. Σας ευχαριστούμε κυρία Κάντεμπαχ. Φυσικά θα επανεμφανιστεί στην εμείς διάταξη αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Σας συγχαίρουμε και σίγουρα δεν έχουμε κάθε μέρα τέτοια τέτοιες εκθέσεις για ένα τόσο ε, συγκεκριμένο ζήτημα και τόσο σημαντικό ζήτημα. Θέλετε, κύριε Γέμπερ, ε, να κάνετε καταληκτικές παρατηρήσεις. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μόνο μια σύντομη παρατήρηση. Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχεται την ουσία των συστασιών μας. Και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα υλοποιηθούν. Πάντως, όπως ε, είπαμε στην εκθεσή μας είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι η σχέση μεταξύ της υπαίθρου και των στόχων των νέων πηγών ενέργειας. Ακόμη το 95% των πόρων υπάρχουν και θα πρέπει να αξιοποιηθούν για ανάπτυξη της υπαίθρου και όχι σε επιλεγμένους γεωργούς. Επίσης να σας πω για την δεύτερη οδηγία για ανανεώσιμη ενέργεια είπαμε ότι υπάρχει τώρα διεκλογία φιλεγραδών μελών αλλά υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι από αυτή την πρόταση κάποιοι κίνδυνοι που έχουν σχέση με την εντατικοποίηση της γεωργίας, διαχείριση των δασών εκπομπές δηλαδή κάποιων ρηπαντικών μολυσματικών ουσιών σε σχέση με τόσο προβλέπει η οδηγία. Άρα θα πρέπει όταν έρθει η ώρα έγκρισης της οδηγίας να ληφθούν και αυτοί οι υπόψη. Ε, ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε την σύντομη παρουσίαση αυτής της έκθεσης και περνάμε στην επόμενη έκθεση. Συγκεκριμένα την υπαρισμό 10 ε, το σύστημα βασικών πληρωμών για τους ε, γεωργούς. Ε, η κυρία Σμίτ από, την, από το Ελληνικό Συνέδριο είναι η αρμόδια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. of Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι τιμή μου, κύριοι βουλευτές, με αυτή την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τα βασικά συμπεράσματα αυτό του οικονομικό ελέγχου όσον αφορά ε, αυτό το πρόγραμμα, το πλαίσιο πληρωμών για τους αγρότες. Ελπίζουμε ότι έτσι θα είναι καλύτερη επικοινωνία και αυτό το βασικό σύστημα πληρωμών εγκρίθηκε στην μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 13 και αντικατέστησε το SPS και είπαμε να προβλέψουμε πληρωμές στους γεωργούς επί τη βάση αυτού του πλαισίου. Και όπως ξέρετε το SPS αφορούσε την αποσύνδεση και οι γεωργοί ε, ε δίκαιωσαν κάποιες ε, πληρωμές επί τη βάση της επιλέξιμης γης που κατήχαν. Όπως ξέρετε αυτό αφορά κάποια αιτήσια έξοδα για περίπου 18 δις ευρώ και αφορούσαν 4 εκατομμύρια αγρότες σε 18 χώρες μέλη και ε, η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη συνδιαχειριζόντουσαν το σύστημα BPS. Σημασία του οικονομικού ελέγχου είναι το ότι είναι ως σύστημα αυτό λειτουργικό, αλλά έχει περιορισμένες επιπτώσεις όσον αφορά την απλούστευση, το targeting και την κάλυψη 8 επιπέδων. Τι άλλα συμπεράσματα έχουμε. Στον τον υπολογισμό της χρέωσης, εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι αρχές των καταβολών των κρατών μελών θα πρέπει να κάνουν σημαντικές προσπάθειες και σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε μόνο υπολογισμό προσωρινό και κάποιες υπηρεσίες πληρωμής είχαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Αλλά τονίζουμε ότι οι πληρωμές του συστήματος BPS γενικώ δεν έπασχαν από σφάλματα. Τώρα, όσον αφορά την διαχείριση του BPS, καταλήξαμε στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε αρκετές ε, οδηγίες στα κράτη-μέλη, αλλά δεν μπόρεσε πάντοτε να εξασφαλίσει την συνεπή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Όσον αφορά τώρα την απλούστευση, σας συμμεθυμίζουμε ότι αυτή ήταν μία από τις αρχές της μεταρρύθμισης του 2013 και η περίπλοκη κανόνες της Ένωσης για το BPS και την επιλέξιμη γη περίχαν πάρα πολλές εξαιρέσεις για την εφαρμογή αυτού του πλαισίου και οι επιλογές που είχαν τα κρατημέλη δεν ήταν πάντοτε υπέρ της απλούστευσης. Πολλές φορές προσέθεταν πολυπλοκότητα. Όσον αφορά τώρα την στόχοθέτηση, το targeting, καταλήξαμε στο ότι αυτή η μεταρρυθμίση επίσης και τις κατηγορίες για τη γη και όπου υπάρχει κάποιο είδους ε, στήριξη, σχετικέ πληρωμέ δηλαδή, και απαιτείται μια ελαχίστη γεωργική δραστηριότητα. Για κάποια κράτη-μέλη ε, υπήρχε κάποια μερική εφαρμογή του προγράμματος και σε κάποια μέλη υπήρχε κάποια δυναμική ε, προσέγγιση ούτω ώστε είχαμε κάποιο είδους αρνητικές συνέπειες, δηλαδή κάποιο είδους ε, παράνομες αξιώσεις και μετά η, το επίπεδο στήριξη σε ένα εκτάριο απέκτησε περισσότερη ομοιογένεια αλλά σε 11 κρατη από τα 18 έχουμε συνδέει σημαντική διαφορά που θα μετά το 2019. Γι' αυτό και καταλήξαμε ότι το BPC έχει σημαντικά όρια, περιορισμούς όσον αφορά το να καλύψει τα προβλήματα εισοδημάτων των γεωργών και τελικά είναι υπέρ των μεγάλων, των μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων. Και επίσης το ότι δεν υπάρχουν σαφείς ε, στόχοι και κατά κάποιο τρόπο μια σταθερή αφετηρία κάνει το σύστημα λίγο αποτελεσματικό και επίσης δεν προσφέρει το σύστημα αρκετή προστήριξη. Οπότε, επί τη βάση όλων αυτών συστήνουμε να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα θα πρέπει να καλύψουν αυτέ τι αδυναμίες ε, όσον αφορά κάποιου σημαντικούς ελέγχους και να διορθώσουν ε, τα σημεία στα οποία οι τιμές επηρεάζονται από την μη εφαρμογή των σχετικών κανόνων και για το ότι δεν υπάρχει επικαιροποιημένη ε, ενημέρωση, δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη χρήση της γης επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεπής ερμηνεία και εφαρμογή του νομικού πλαισίου για το σύστημα BPS επίσης. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση της ισχύου νομοθεσίας ούτως ώστε να εφαρμοστούν σημαντικές πληροφορίες που αφορούν ε, τα προγράμματα άμεσης στήριξης. Επίσης θα πρέπει οι οργανισμοί επιστοποίησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δουν το κατά πόσο υπάρχουν κατάλληλοι έλεγχοι όσον αφορά το ποιοι θεωρούνται ε, ε, επιλέξιμοι για το BPS και να υπάρχουν ακριβείς υπολογισμοί για το σύστημα. Και θα πρέπει επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν προβήσει οποιαδήποτε πρόταση για την μέλουσα χάραξη και διαμόρφωση της ε, ΚΑΠ να αναλύσει τις ε, ανάγκες του εισοδήματος για κάθε ομάδα γεωργών και να δει ποια, ε, ποιοι είναι οι λειτουργικοί στόχοι οποιοδήποτε μηχανισμού του εισοδήματος και να δει πώς είναι δυνατόν να επιτεθούν αυτοί οι στόχοι και να συνδέσει αυτές τις εξαρχές από την μέτρα σε κάποιο είδους ενδεδειγμένους λειτουργικούς στόχους και αφετηρία ενεργειών, ούτω ώστε να είναι δυνατόν να υπάρχει συγκρισιμότητα για το πόσο αποδίδει η στήριξη του εισοδήματο. Οπότε γι' αυτό και καταλήξαμε ότι ε, τελικά αυτά προτείνουμε θα τα δεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε το ίδιο μήκο κύματο νομίζω ότι βέβαια υπάρχουν και δυσκολίε διότι περιμένουμε νέε προτάσει για την νέα ε, περίοδο της ΚΑΠ, για την περίοδο δηλαδή μετά το 2020. Όταν το οικονομικό έλεγχο εκεί καταλήξαμε και ε, σας είπαμε ποιες είναι οι συστάσεις που έχουμε διατυπώσει και είμαστε στην ε, διάθεσή σας να βάλετε τις ερωτήσει που έχετε και σας ευχαριστώ. Πρόεδρε. Fragen ευχαριστούμε. Η κυρία Σμίτ είναι η συγγετρία μας, παρακαλώ. Με ναι, ευχαριστώ για την έκθεση. Δυστυχώς, ξέρουμε ε, όταν παίρνουμε μια τέτοια ειδική έκθεση ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει η μεταρρύθμιση, δεν θα είναι μετρήσιμη η στόχη, γιατί είναι υπερβολικά μεγάλες οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ξέρουμε ότι οι εθνικές αρχές επίσης επιβαρύνονται με ε, ε, υπερβολική γραφειοκρατία και άρα αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Μέσα στην έκθεση βρήκα, θέλω να παραθέσω κάτι από μία Την έκθεση που ε, συνοψίζει την έκθεση λέει «Ο στόχος της συνθήκης είναι να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη της υπαίθρου και βιώσουμε σε συνθήκες διαβίωσης ε, καθώς και την, ε, το παρκές γεωργικό εισόδημα. Αυτοί οι στόχοι δεν έχουν όμως προσδιοριστεί επακριβώς και δεν έχουν μεταφραστεί σε μετρήσιμα κριτήρια και άρα δεν υπάρχει απόδειξη για την αποτελεσματικότητα της επιδότησης σε σχέση με την εξασφάλιση ε, βασικού γεωργικού εισοδήματος. Βλέπουμε λοιπόν Ποιο είναι ε, το πιο αποτελεσματικό, ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να χρησιμοποιήσουμε τις γεωργικές ενισχύσεις για να στηρίξουμε την παραγωγή γεωργικού εισοδήματος και για να έχουμε μετρήσιμους στόχους. Εγώ θα ήθελα να στηρίξουμε τους στόχους της, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά οφείλω να πω ότι δεν συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό του ελεγκτικού συνεδρίου, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τι ωραία ενέκρινε κάποιες συστάσεις, μα θα έπρεπε ούτως ή άλλως να τις εγκρίνει ε, και Συμφωνώ απολύτως λοιπόν με την άποψη και τους στόχους του ελεγκτικού συνεδρίου και θεωρώ ότι θα πρέπει να λειτουργεί ικανοποιητικά το σύστημα ελέγχου παρά το γραφειοκρατικό άχθος που αυτό συνεπάγεται. Για όποια ε, κράτη και αν μιλάμε, ε, για τη Γεωργία, για τη Σουηδία, για την Πορτογαλία, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται με ομοιόμορφο τρόπο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι τα καθήκοντα που θα αναλάβει εκείνη και ποια καθήκοντα αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη, ώστε ε, να ε, ελέγχουμε την, αποτελεσματικά την ε, καταβολή των πληρωμών για τις γεωργικές αξιώσεις. Μόλις γνωρίζουμε και τα ποσά για τη μελλοντική γεωργική πολιτική θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι αλλά φυσικά δεν θα πρέπει να στηρίζουμε μόνο τους δικαιούχους αλλά και την γεωργική παραγωγή για την ε, ε, εξεργασία τώρα αυτής της ε, ειδική έκθεσης φυσικά παραμένουμε ανοιχτοί και θέλουμε όπως είπαμε να εκπροσωπούμε και τα συμφέροντα του γεωργού, γεωργού του φορολογουμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ομοιόμορφο τρόπο. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα εγκρίνει μόνο κάποιες προτάσεις και συστάσεις, αλλά ευελπιστώ ότι θα εγκρίνει όλες τις συστάσεις του ελληνικού Συνέδριου. Εμείς είμαστε υπερ. Ευχαριστούμε κυρία αν κατάλαβα καλά η βασική και σημαντική σύσταση είναι υπαριθμόν 3. Ένα νέο νομικό πλαίσιο που θα προσδιοριστεί μετά την ανάλυση των επιπτώσεων του προηγούμενου πλαισίου. Δηλαδή ποιο θα παίρνει τα λεφτά και για ποια πράγματα ε, υπάρχουν τα λεφτά, αλλά γι' αυτό δεν ξέρουμε τίποτα γιατί από ό,τι κατάλαβα το Μάιο μόνο θα έρθει ε, η πρόταση νομοθετικού περιεχομένου, οπότε μήπως θα έπρεπε να τα πάρουμε με τη σειρά και ε, αυτή, θα, αυτή η πρόταση θα είναι και η βάση ούτως ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερες επενδύσεις σε μεγαλύτερα γεωργικά ε, τεμάχια. Ο Διευθυντής Μπάσκο και ο αναπληρωτής Διευθυντής από την Γενική Διεύθυνση. Ποιος θα πάρει το λόγο έχουμε και τους δύο εδώ πέρα. Σύντομη παρουσίαση θα κάνουμε. Ούτως ή άλλως ε, δεν θα ολοκληρώσουμε σήμερα. Διεξοδικότατα και μελλοντικά θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα. Δεν θέλουμε θύμα, θέλουμε κάποιον που να υποστηρίζει τις απόψεις του. Αποφασίστε το μεταξύ σας. Ε, λοιπόν, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, ε, ευκαιρία που μας δίνει να, κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για την ελληνική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για το σύστημα πληρωμών. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για την έκθεση και όλες οι συστάσεις που έχουν ε, ειδικό βάρος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίθηκαν όλες και θέλω να επιμείνω και να το τονίσω αυτό. Θα δούμε τώρα μέσα στις προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου που τώρα εξετάζονται και προετοιμάζονται για την περίοδο μετά το 2020 θα συμπεριλάβουν αυτές οι συστάσεις. Αναγνωρίζουμε ότι ε, έχει εγκριθεί το βασικό σύστημα πλογών και παρακολουθούμε την ε, εφαρμογή του, παρέχουμε σε γραμμέ και είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα. Και τώρα θέλω να τονίσω πώ είναι πολύ σημαντική αυτή ε, σημαντικό αυτό το συμπέρασμά σας για το βασικό σύστημα ε, πληρωμών για τους γεωργού. Επίσης, ε, το συμπέρασμά σας για την εισαγωγή του EPS που συνεπάγεται πολύ σημαντικές προσπάθειες από τα κράτη-μέλη αλλά και από τις αρμόδιες αρχές. Πολύ θετική αυτή η σύσταση, όμως είναι φυσιολογικό. Επειδή είναι περίπλοκη διαδικασία να υπάρχουν και λήψεις. Και εδώ αναθεώρησαν οι ελεγκτές την δουλειά των κρατών μελών και Συνεχίζονται οι έρευνε ώστε να προστατευτεί ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι επιχειρησιακώ πώ ακολουθούνται ε, τα όσα είχαν προβλεφθεί, όμω χρειάζεται απλούστευση του συστήματο και δεν έχουν γίνει επαρκεί προσπάθειε για τη σύγκληση των στόχων. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι ενώ στην αρχική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαμε λιγότερε εναλλακτικέ λύσει και ήταν πιο απλό το πρόγραμμα, αληθεύει ότι ε, στα πλαίσια τη ε, συνομοθετική ε, διαδικασία για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ αναγνωρίζεται ότι θα πρέπει να χορηγηθεί μεγαλύτερο περιθώριο λιγμονών στα κράτη-μέλη, αλλά αυτό οδηγεί δυστυχώ και σε πιο περίπλοκους κανόνες. Σε σχέση με τη στόχευση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να στοχεύσουν την υποστήριξη προς τους ενεργούς γεωργούς και θα πρέπει να διαφοροποιήσουν ενδεχομένω τη βασική πληρωμή για δύο διαφορετικά καθεστώτα Ξέρουμε ότι για την περίοδο μετά το 2020 έχουμε εξαγγείλει στην τελευταία ανακοίνωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε την επιθυμία της να υποστηρίξει τους πραγματικούς γεωργούς, δηλαδή αυτοί που ενεργά ε, ακολουθούν αυτή την εμπορική δραστηριότητα για να εξασφαλίσουν τα ζήτημα. για τη σύγκληση. Τρει εναλλακτικέ λύσει για την εσωτερική σύγκληση. Πρώτη για την πλήρη σύγκληση βραχυπρόθεσμα. Ε, μία δεύτερη για την πλήρη σύγκληση ή μεσοπρόθεσμα και μια για μερική σύγκληση για το εσωτερικό μοντέλο όπως το ονομάζουμε που θα επηρεάσει ε, τις, τα αποτελέσματα αυτής της ε, εφαρμογής του καθεστώτος από τα κράτη-μέλη όμως εκεί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές από κράτος σε κράτος και θέλω να τονίσω ότι η εφαρμογή της περιφερειοποίησης δηλαδή η διαφοροποίηση των πληρωμών ε, έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του βαθμού της σύγκλησης ανά κράτος μέλος. Επιπροσθέτω, το ελεγκτικό συνέδριο τονίζει ότι το τωρινό σύστημα δεν βασίζεται στη συνολική κατάσταση του γεωργικού εισοδήματο και θέλω να τονίσω εδώ πω Θέλουμε να επιθυμήσουμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική εξασφαλίζει τη στήριξη εισοδήματο μέσω τη στήριξη γεωργική δραστηριότητα. Δηλαδή, ενθαρρύνουμε του γεωργού να έχουν ε, τακτική γεωργική δραστηριότητα και αυτό συνάδει με τη συνθήκη. Μέσα σε αυτό το σύστημα βασικών πληρωμών, λοιπόν, ε, εστιάζουμε ε, στο εισόδημα που προέρχεται από αυτέ τι γεωργικέ δραστηριότητε, και από την ε, τους ε, ε, παράγοντες παραγωγής, δηλαδή μέτρα δεύτερου πυλών όπως παραδείγματος χάρη δραστηριότητες διαφοροποίησης, όπως ο αγροτουρισμός. Λοιπόν, η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της γεωργίας και της διατροφικής πολιτικής από τον Νοέμβριο 2017 προτείνει για την επόμενη προγραμματική περίοδο μεγαλύτερη επικουρικότητα ε, και ένα νέο σύστημα για το σύστημα, ε, ε, μία νέα μέθοδο για το σύστημα EPS ε, ε, ESP, συγγνώμη, ε, όπου τα κράτη-μέλη θα έχουν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών, αλλά θα είναι και πιο υπόλογα για την επίτευξη των στόχων, για την εξαγωγή των ελέγχων και πώς θα συνδέονται δραστηριότητε με ένα στρατηγικό σχέδιο. Η πρότασή μας θα λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία που έχουμε για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής του Στήματος πληρωμών και θα εξετάσουμε διεξοδικά όλα αυτά τα στοιχεία, κυρίως αυτό τη στήριξη, διότι για να έχουμε μια ομοιόμορφη κατανομή τη στήριξη ανάμεσα στους δικαιούχους ε, τη κοινή γεωργικής πολιτική είναι από τους βασικότερους στόχους της μελλοντικής γεωργικής πολιτικής και σε αυτή το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει πώς θα στοχεύσουμε την παραγωγή του εισοδήματο, αλλά όχι μόνο ανά μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευση, αλλά και ανά είδος ε, ε, ε, ε, και, το εισόδημα δεν προέρχεται μόνο από γεωργική δραστηριότητα, αλλά όπως είπα και από εναλλακτικές πηγές, όπως διαφοροποίηση γεωργικής δραστηριότητας. Ευχαριστώ. Ναι, δεν κατάλαβα τι κάνουμε εδώ. Δεν το κατάλαβα, λυπούμε πολύ. Θα πρέπει να μου το πείτε και πάλι. Ποιο είναι το πλάνο αυτή τη στιγμή. Η έκθεση είναι μια θεμελιώδης κριτική ε, για την πολλωστή φορά στο σύστημα. Για πείτε μου τα βήματα, το πώς η Επιτροπή θέλει να προσεγγίσει μία ανάλυση του ερωτήματος κατά πόσο θέλουμε να κάνουμε τους πλούσιους πλουσιότερους, τους μεγάλους μεγαλύτερους μέσω του συστήματος ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Είχαμε πάει στην ε, Τσεχοσλοβακία θα επανέλθουμε εδώ και πραγματικά θέλουμε τη δική σας ε, πραγματογνωμοσύνη. Πείτε μας με απλά λόγια τι μπορούμε να περιμένουμε όσον αφορά τις αναλύσεις και τις επισημάνσεις για το θέμα αυτό. Και κατ' εξαίρεση θα δώσω προηγουμένως το λόγο σε δύο συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, συγγνώμη αν ε, παρανόησα. Ε, καταρχήν θα ήθελα να διευκρινίσω. Αλλά αυτή η έκθεση δεν μιλάω για τι συστάσει, αλλά για τα συμπεράσματα και την ουσία των παρατηρήσεων που είναι κατ' ουσίαν θετικέ όσον αφορά την εφαρμογή του βασικού σχήματο πληρωμών και διευκρινίζει κάποια θέματα όσον αφορά τι ελλείψει στη στόχευση, την περαιτέρω ανάγκη απλούστευση και και διάφορα θέματα που αφορούν τη σύγκληση. Ε, όσον αφορά την κάθε χώρα μέλος. Αυτές είναι, αυτή είναι η βασική στόχη που έχουμε να ε, προσεγγίσουμε μελλοντικά στο επίπεδο τη ε, κοινή ε, γεωργική πολιτική. Το περασμένο Νοέμβριο στην ανακοίνωσή μα, ε, τονίσαμε ότι επιθυμούμε να υπάρξει μια απλούστευση τη κοινή γεωργική πολιτική, ένα εξυγχρονισμό, ούτως ώστε να πετύχουμε του στόχου μα, επίση αύξηση του βαθμού δικαιοσύνη, όσον αφορά την επιτεύξη των στόχων μα και, θα ήθελα και επίση θέλουμε να αναφέρουμε κάποιε άλλε σκέψει εν σχέση με δυνατότητε εισαγωγή κάποιων κατοφλίων ή διαβάθμισης των ε, πληρωμών ένας καλύτερος συστήματος διανομής ε, ε, προς γεωργούς οι οποίοι εξαρτώνται από αυτή τη δραστηριότητα όσον αφορά τη διαβίωσή τους. Επίσης επιθυμούμε να εφαρμόσουμε ένα νέο σύστημα για την γεωργική πολιτική, το οποίο θα βασίζεται σε μεγαλύτερη επικουρικότητα, ούτως ώστε να υπάρξει μια νέα ισορροπία ε, ευθυνών μεταξύ ενωσιακού επίπεδου, και επίπεδου των χωρών μελών. Και επίσης θέλουμε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή της, τον και την εφαρμογή της πολιτικής και ε, θα προσπαθήσουμε να παράσχουμε μια βιώσιμη ενίσχυση προς τους ε, γεωργούς και να το συνδέσουμε με την ε, ε, κοινωνική ενίσχυση. Είναι ξεκάθαρο και το είπα ήδη στην εισαγωγή της ομιλίας μου εάν η Επιτροπή αποδεχτεί τις συστάσεις δεν μπορεί να εξετάσει το αποτέλεσμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της ε, νομοθετικής πρότασης. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος ε, Φλέμιγκερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω κάποιους καλλιεργητές από τη δική μου περιοχή και ξέρω τι θα έλεγαν ότι οι πλούσιοι γίνονται με τον τρόπο αυτό πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Αυτό θα έλεγαν. Το πρόβλημα είναι ότι από όσο είμαι σε θέση να κατανοήσω ε, θα μπορούσαμε να προβούμε σε απλούστερες λύσεις και να εγγυηθούμε, να εγγυηθούμε ότι τα χρήματα πηγαίνουν στους μικρούς καλλιεργητές. Εάν είχαμε μικρότερη, λιγότερη επικουρικότητα από ό,τι εδώ. Αλλά βρισκόμαστε ε, σε μία κατάσταση όπου ένας καλλιεργητής μπορεί να πάρει 1000 ευρώ για ένα εκτάριο και ο διπλανός καλλιεργητής να πάρει 60 ευρώ. Ε, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αν έχουμε περισσότερη επικουρικότητα, τι θα γίνει σε μέρες κλοκές περιφέρειε, για παράδειγμα στη δική μου, όπου υπάρχει τεράστια, ασκείται τεράστια πίεση για να μην υπάρξουν αλλαγές. Ε, πώς ε, θα γίνουν αυτές οι αλλαγές ε, υπό το πρίσμα της μεγαλύτερης επικορικότητας των πυλώνα 1. Ε, το σύστημα αυτό είναι εξαιρετικά... Και τι γίνεται με τον πυλώνα 2. Είναι εξαιρετικά πολύπλοκο το σύστημα. Και αν ε, κάνουμε όπως στην Ιρλανδία, όπου λαμβάνεται η απόφαση ε, και λέγεται ότι αν πληρούνται αυτά τα κριτήρια, έχει καλός. Τι έγινε και με τον πυλώνα 2 στο παρελθόν. Νομίζω ότι πραγματικά είναι γελιοδός ε, πολύπλοκο όλο αυτό το σύστημα. Ε, δεν βλέπω πώς ε, θα απλουστευτεί το σύστημα αυτό και πώς θα εγγυθούμε τις ροές χρημάτων προς καλλιεργητές. Γιατί πιστεύω ότι ε, αν είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε τις αποφάσεις στις περιοχές μας τότε όταν ερχόμαστε μας έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να ανισχύουμε πλέον τους μικρούς καλλιεργητές γιατί δεν υφίστανται. Ε, ναι. Η κυρία Χόιμπουχ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Με απελπίζει όταν ε, θέλουμε απλούστευση ε, και στόχευση. Ε, όσον αφορά τις βασικές ε, ενισχύσεις ε, εννοούμε το, ίδια, το ίδιο ποσό για το ίδιο εκτάριο. τότε δεν υπάρχει καμία στοχοθεσία και το αποτέλεσμα είναι ότι οι πλούσιοι γίνονται πλησιότεροι ενώ οι φτωχοί προσπαθούν να επιβιώσουν. Όταν μιλούμε για επικορικότητα λέμε ότι θα αφήσουμε περιθώριες στις μέλη να δουν πώς θα πετύχουν ε, κάποιους στόχους. Ναι, ωραία, αλλά μόνο εφόσον είναι ξεκάθαρα, υπάρχει ένας ξεκάθαρος ορισμός των στόχων, οι οποίοι είναι ανεπαρκώς, ε, ε δεν είναι αρκετά ξεκάθαροι. Ε, όσον αφορά τους ε, περιβαλλοντικούς στόχους και λοιπά, την κλιματική αλλαγή. Ε, εδώ υπάρχει μεγάλη ασάφεια και θα πρέπει να αποφασίσουμε τι δυσιοργία επιθυμούμε, τι είναι κοινωνικά βιώσιμο, τι είναι αυτό το οποίο προωθεί το περιβάλλον, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να σταματήσει την κλιματική αναστροφή. Και στη συνέχεια μπορούμε να δούμε ποια εργαλεία είναι τα ενδεδειγμένα. Αλλά να μιλάμε μόνο για απλούστευση και αυτό να το καθορίσουμε εστιάσουμε μόνο στο πλαίσιο μια συγκεκριμένη στόχευση, νομίζω ότι δεν θα μα κάνει να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με του καλλιεργητέ και για, ε, γιατί σε κάθε χώρα μέλο ισχύουν άλλε προποθέσει εντελώ ε, διαφορετικέ. Ε, νομίζω ότι τα κατόφλια και η, μια διαβάθμιση προς τα κάτω θα ήταν ίσως κάποιες ε, δυνατότητες αλλά πρέπει να είμαστε πολύ πιο ξεκάθαρες προς τους στόχους και να δούμε πού ακριβώς πάνε τα χρήματα. Απλούστευση και στόχευση ταυτόχρονα νομίζω ότι δεν είναι εφικτό. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και το ελληνικό συνέδριο. Από όλη αυτή τη συζήτηση για την ΚΑΠ. Αυτό το οποίο λείπει είναι να ακούσουμε τη γνώμη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, είμαστε εδώ συνομοθέτε. Και ο Λένα και πιο μεγάλο κάνουμε το στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Παρ' όλα αυτά, να τα τώρα τα προβλήματα. Ε, να δούμε βέβαια τι θα κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και σα λέω ότι θα ήθελα αυτέ οι συστάσει να αξιοποιηθούν και εδώ και στο Συμβούλιο με περισσότερες υποχρεώσει γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική να αποδώσει στο μέλλον και να ωφεληθούν οι ευρωλογούμενοι. Είναι θεμητό να το θέλουν αυτό. Το ναι, δηλαδή αποτελεσματική κάποια να κάνει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Τώρα, πρώτο αφορά το ελληνικό συνέδριο. Εντάξει, δύσκολο είναι, αλλά πετε μα δύο λόγια. Τι είναι, νομίζετε, όσον αφορά την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον των ε, τροφίμων για τις ε, γεωργίε, τι γίνεται για τι ε, συζητήσει που θα ακολουθήσουν, τι διαπραγματεύσει που θα ακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή και μετά το ελεγκτικό συνέδριο. Thank you, Mrs. Chair. Σας ευχαριστώ να επανέλθω πρόεδρε σε κάτι, κάτι το οποίο αναφέρθηκε όσον αφορά τη στοχοθέτηση, την ε, απλούστευση, την ε, επικουρικότητα. Ε, βέβαια, είναι βασικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να τονιστεί στην ε, ανακοίνωση τέλους Νοεμβρίου. Στο μέλλον δηλαδή, είτε η γενική είτε η ειδική λειτουργική στόχη της ΚΑΠ στήριξη, ανθεκτικότητα, ευφύς, αντιμετώπιση κλπ. κλπ. Για να λύγει το κλίματος ακόμα θα πρέπει όλα αυτά να είναι πιο σαφή. Και αυτή η σαφή στόχη θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε εθνικό επίπεδο που να έχουμε κάποιο είδους ποσοτικά αποτιμόμενα στοιχεία και αποτελέσματα από τα κράτη-μέλη για το πώς θα επιτευχθούν αυτή η συγκεκριμένη στόχη. Να λειτουργεί περισσότερο η επικουρικότητα όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών στα κρατη για το πώς θα επιλεχθούν αυτοί οι λειτουργικοί συγκεκριμένοι στόχοι. απλούστευση, στοχοθέτηση, σύγκληση. Όλη αυτή η θα πρέπει στο μέλλον να έχει βάση ένα στρατηγικό πρόγραμμα. Και να μας λένε τα κρατημέλη τι θα κάνουμε με την, ε, ε την κρατική παρέμβαση. Βέβαια, να μην ξεχνούμε ότι όσο περισσότερους στόχους βάζουμε, τόσο περισσότερες προϋποθέσεις ε, θέτουμε και για την επιλεξιμότητα κλπ. Θα σπίσουμε περισσότερες προϋποθέσεις για να δοθούν τα προβλεπόμενα ποσά στους ε, επιλέξιμους, στους δικαιούχους τέλος πάντων. Ε, δύσκολο να βρει κανείς σωστή η ισορροπία μεταξύ καλύτερη στοχοδέτησης και περισσότερη απλούστευση. Ε. αυτά κάνει η σημερινή ΚΑΠ για το πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Πριν από μερικές εβδομάδε μιλήσαμε για το πράσινισμα και λέμε και ότι και τώρα σε εθνικό επίπεδο ίσως οδηγηθούμε σε περισσότερη περιπλοκότητα σε κάποιες χώρες. Αυτό θα πρέπει στο μέλλον να το αντιμετωπίσουμε με τα στατικά προγράμματα, κάποια διαδικασία διαρθρωμένη, με επικουρικότητα των πρώτων μελών, βελτίωση στοχοθέτηση και να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις όσον αφορά τη γραφειοκρατία. Also, für uns Ausschuss wird es bedeuten... Για τη δική αυτό θα σήμαινε ότι θα πρέπει να παλέψουμε με 25, 27 διαφορετικά συστήματα. Πώς ο καθένας κάνει τι και το ίδιο θα πρέπει να κάνει και το ελεγκτικό συνέδριο, πράγμα που θα ήταν εξαιρετικά προβληματικό προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα η Επιτροπή Γεωργίας να δέχεται ακόμα περισσότερες πιέσεις από ό,τι στο παρελθόν, γιατί υπάρχουν χώρες ε, μέλη όπου υπάρχουν ε, κάποιοι πλούσιοι στην κυβέρνηση, όσον αφορά στη Σλοβακία για παράδειγμα. Ε, και δεν υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και πολλά ερωτηματικά όσον αφορά το σύστημα της Βουλγαρίας ε, και με τον τρόπο αυτό θα ανοίξουν όλες οι πόρτες, οι ασκή του αιώλου. Και έχω σημαντικές αμφιβολίες εδώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας αρέσουν οι προκλήσεις και δεν θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Όχι, αντιθέτως. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που θέσατε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Κατά την άποψή μου, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω ότι όλες αυτά, όλα αυτά τα θέματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Γιατί όπως είπε η κυρία Πρόεδρος, πρόκειται για μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Γιατί πράγματι υπάρχουν διαφορετικές αξίες που ορισμένε φορές είναι αντιφαρικές μεταξύ τους και είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε τη σωστή ισορροπία με πολιτικούς όρους. Καταρχήν, θα ήθελα να πω το εξή. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου, η μη ικανοποίησή μου, για το γεγονό ότι οι συστάσει δεν έγιναν όλε αποδεκτέ. Βεβαίω, θα ήμουν πιο ικανοποιημένο εάν είχαν γίνει αποδεκτέ όλες οι συστάσεις. And I must say also... Θα πρέπει να πω επίσης ότι πιστεύω ε, τις στάσεις αυτές και γι' αυτό έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο. Ακόμα ε, και γνωρίζοντας ότι η Επιτροπή δεν συμφωνεί με όλες αυτές. Εμείς όμως θεωρούμε ότι όλες αυτές οι στάσεις είναι σημαντικές και θα έπρεπε να συμπεριληφθούν, να διατηρηθούν στο κείμενο, έστω και συνοδευόμενος από κάποιες κριτικές σκέψεις. Βεβαίως η Επιτροπή βρίσκεται σε μια ευαίσθητη θέση αυτή τη στιγμή γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται η αναθεώρηση ε, της ε, ΚΑΠ η οποία έγινε το 2016 και αυτή τη στιγμή ε, η Επιτροπή ε, προβαίνει σε μια νέα αναθεώρηση άρα ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δύσκολη θέση της. Αλλά όπως σας είπα, όσον αφορά τις σημαντικές, τα σημαντικά θέματα, αυτό το οποίο λέμε στο νομοθέτη είναι το εξή. Όταν εγκρίνατε τη μεταρρύθμιση το 2013 και γνωρίζουμε ότι αποτέλεσε τον καρπό μακρών συζητήσεων ορισμένοι από τους βασικούς στόχους τους οποίους εσείς επισημάνατε όπως είναι η απλούστευση η, σύγκληση των ε, λύσεων ε, διαπιστώσαμε ότι ε, δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν. Και το λεκτικό Συνέδριο έχει την υποχρέωση να αναφέρει στο νομοθέτη τα προβλήματα όσον αφορά την ε, απλούστευση. Εδώ εφίστανται κάποια προβλήματα και είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξουν προβλήματα μεταξύ ε, επικουρικότητας και ανάγκης απλούστευσης. Εμείς ε, διαπιστώσαμε επίσης κάποια προβλήματα όσον αφορά τη στοχοθέτηση. Στην ε, αναθεώρηση 2013 εισήχθη η έννοια των ενεργών ε, καλλιεργητών προκειμένου να δοθεί ενίσχυση προς τους πραγματικούς ε, αγρότες, γεωργούς. Γιατί και ακριβώς διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν προβλήματα όμως στην εφαρμογή αυτού του μοντέλου. Επίσης όσον αφορά τη σύγκληση και εδώ διαπιστώθηκαν ε, προβλήματα. Ήταν ε, μια από τις, ένας από τους βασικούς ε, στόχους της του 2013 η σύγκληση και πιστεύω ότι θα υπάρξουν διαφορές και μετά το 19 και αναγνωρίζουμε ότι τελικά το σύστημα αυτό κατατείνει να ευνοεί τους μεγάλους καλλιεργητές. Και αυτό μας φέρνει στο θέμα το οποίο συζητήσαμε πριν από λίγο σε σχέση με τα έσοδα και τη στήριξη των εισοδημάτων των γεωργών. Γιατί στο τομέα αυτό εγώ πραγματικά κατανοώ την θέση της Επιτροπής, αλλά πιστεύω ότι γνωρίζοντας τις δυσκολίες, γιατί βεβαίως υφίστανται δυσκολίες, δεν είναι εύκολη αυτή η υπόθεση, λέω ότι δεν θα έπρεπε να δηλώσουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι ε, γνωρίζοντας μόνο τα έσοδα τα οποία παράγονται από τις, ε, δραστηριότητες, από τις γεωργικές δραστηριότητες. Γι' αυτό διατυπώσαμε τη σύσταση παριθμών 3, όπου λέμε ότι η ενίσχυση των εισοδημάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την τον τρέχοντα επιμερισμό της ε, ενίσχυσης που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων περιοχών, το κόστος και την ε, ποικιλότητα των τρόπων ε, καλλιέργειας. Και θα ήθελα να ζήσω από τον νομοθέτη πραγματικά να στρέψει την προσοχή του προς τον τομέα αυτό, γιατί φοβούμαι ότι αν ε, δεν ε, προσέξουμε όλα αυτά τα θέματα, προσπαθώντας ε, να πετύχουμε μια νέα στοχοθέτηση της νέας ΚΑΠ, θα αποτύχουμε. Και τέλος, ε, λαμβάνοντας υπόψη μου τις ερωτήσεις που τέθηκαν, θα έλεγα το εξής. Εμείς εδώ συζητούμε μόνο το βασικό, το BPS, το βασικό μοντέλο πληρωμών για τους ε, γεωργούς το οποίο σχετίζεται όμως συνάρτητα με τη μελλοντική διαφόρμωση της ΚΑΠ και πιστεύω ότι το θέμα αυτό τελικά θα καταλήξει το εξής το κατά πόσο το ελεγκτικό συνέδριο ε, θα μείνει στη θέση του όσον αφορά τη μελλοντική διαμόρφωση της ΚΑΠ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει η συγγήτρια να πάρει το λόγο. Καταληκτικά όχι. Τότε ε, νομίζω θα πρέπει να συζητήσουμε μελλοντικά το θέμα αυτό διεξοδικά και τότε θα πρέπει να που βάλει και μια αναφορά η Επιτροπή. Ε, Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και ερχόμαστε στην ε, έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για το μέλλον της ΚΑΠ. Η είναι ο κύριος Τσέλερ. Παρακαλώ. Thank you, ε, Chairman. Chairwoman. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, θα ήθελα εν συντομία να σας ε, παρουσιάσω αυτό το ε, ενημερωτικό την ε, ενημερωτική παρουσίαση για να τροφοδοτήσω τις συζητήσεις σας. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας υπενθυμίσω, αν και το γνωρίζετε, ότι έχει εκδώσει ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον ε, των τροφών και της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως απόκριση της Επιτροπής ε, στην ειδική εκθέση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ξέρουμε ότι γίνεται μια ευρύτατη συζήτηση για το μέλλον της ε, ΚΑΠ και προγραμματίζοντας το 2018 θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, εκπονήσουμε κι εμείς μια έκθεση για, το, για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον των τροφών και της γεωργίας Και τονίζω, υπογραμμίζω, δεν είναι ε, ε ελεγκτική έκθεση. Είναι έκθεση αναθεώρησης, ε, βασίζεται σε ε, προηγούμενες ανακοινώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε άλλες δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. Λοιπόν, σε αυτό το, ενημερω... σε αυτό το ενημερωτικό έγγραφο Εκτεδάζουμε τρία βασικά σενάρια. εξετάζουμε ποια είναι τα δεδομένα που είναι σημαντικά για τη Γεωργία και για την Ήπεθρο. Βασιζόμαστε σε άλλες σχετικές πηγές ε, δεδομένων και και προσπαθούμε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα της Γεωργίας και της Ήπεθρου. Το πρώτο κομμάτι του εγγράφου είναι η περιγραφή της κατάστασης της γεωργίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Το δεύτερο τμήμα της έκθεσης είναι τα απορίσματά μας από την ανάλυση της ε, τωρής κοινής γεωργικής πολιτικής. Επισταμένα ε, μελετήσαμε την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε σχετισμό με τις βασικές ιδέες της ανακοίνωσης σας υπενθυμίζουμε εμείς τα προηγούμενα πορίσματα. Τα πορίσματα που συμπεριλάβανε σε προηγούμενα σε προηγούμενες μελέτες και ε, έγγραφα του ελεκτικού συνεδρίου τα περασμένα χρόνια. Και τέλος, ποια είναι τα κριτήρια και ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις μελλοντικής κοινή γεωργικής πολιτικής. Θέλω να τονίσω πως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι πολιτικό όργανο. Δεν έχει αρμοδιότητα για να προσδιορίζει τις ε, ε, πολιτικές... συγγνώμη, το ελεκτικό συνέδριο δεν είναι πολιτικό όργανο. Δεν προσδιορίζει μελλοντικέ πολιτικές. Βάσει της παρελθούσης εμπειρία ε, ως ελεγκτές, εμείς το μόνο που να <coughs> κάνουμε είναι να εισηγηθούμε στον ε, νομοθέτη, όχι τις προτάσεις, μόνο τα κριτήρια για να αξιολογήσει ε, πιθανές προτάσεις στο μέλλον. Αυτή είναι και η πρόθεσή μας στο εν λόγω έγγραφο. Ας δούμε κάποια στάση και κάποια βασικά δεδομένα. Ε, για την, τις δαπάνες που βασίζονται στην στήριξη του εισοδήματος. Και βλέπετε σε αυτό το γράφημα πως ε, εν γέννη η χρηματοδοτική στήριξη στη Γεωργία ε, κινήθηκε σε σταθερά επίπεδο από το 2016 μέχρι το 2018 με διαφορές σε διάφορους τομείς αλλά Εν γέννη, ε, η χρηματοδοτική στήριξη ε, παρέμεινε σταθερά επίπεδα. Δεύτερον, συνοψίζω σε αυτή την πρόταση, λέμε εδώ, λιγότερες αλλά μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, και με μικρότερο φόρτο εργασίας ε, παράγουν μεγαλύτερο output. Οπότε έχουμε υψηλότερο πραγματικό εισόδημα για κάποιον ε, που απασχολείται πλήρως στη γεωργία σε σχέση με το παρελθόν. Πρέπει να ξέρετε πως στην Ευρώπη έχουμε λιγότερους γεωργούς αλλά μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Είναι μικρότερο το εργατικό δυναμικό σε σχέση με το παρελθόν. Και ξέρουμε ότι είναι στα, ε, σταθερή η αξία της, ε, των προϊόντων. Και γι' αυτό ε, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι είναι υψηλότερο το εισόδημα ε, των πλήρως απασχολούμενων στη Γεωργία. Αυτά τα βλέπετε όλα στο γράφημα. Στην ε, ε, πιο σκοτεινή γραμμή ε, είναι ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δεν είναι μειωμένος. Βλέπετε την γραμμή, την κάτω-κάτω γραμμή, είναι τα εισοδήματα αναπλήρως απασχολούμενο που αυξάνονται και στη μέση η γραμμή είναι η προστιθέμενη αξία των προϊόντων η παραγόμενη αξία, αν θέλετε, της γεωργίας που ε, κινείται ε, ε, μάλλον σε σταθερά επίπεδα. Δηλαδή αυξομειώνεται ανάλογα με τη χρονιά, αλλά εν γέννη παραμένει σταθερή η παραγόμενη αξία. Εμείς στο ελεγκτικό συνέδριο θεωρούμε ότι αυτή η γραφική παράσταση ε, συνοψίζει ε, τα, ε, όλα τα πιο σημαντικά δεδομένα της γεωργίας και τις πιο σημαντικές εξελίξεις μέχρι στιγμής. Θέλω να τονίσω κάποια άλλα σημαντικά δεδομένα. Οι τιμέ ε, των τροφίμων, αν κάνουμε μια ε, σύγκριση σε παγκόσμιο επίπεδο και ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, μα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είμαστε καθαροί εξαγωγή τροφίμων, όμω παραμένουμε καθαροί εισαγωγή μη μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων. Η, το, η μέση ηλικία των ε, κατόχων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχει αυξηθεί, αλλά ευθυγραμμίζεται με τις δημογραφικές τάσεις. Ε, τα δεδομένα για την συνολική επιφάνεια εκμετάλλευσης δεν χαρακτηρίζονται από ανακολουθίες, διότι βλέπουμε ότι η συνολική ε, επιφάνεια έχει μειωθεί μέσα από τις στατιστικές για τις συγκομιδές, όμως έχουμε άλλες πηγές που μας δείχνουν ότι το συνολικό εμβαδό έχει παραμείνει σε σταθερά επίπεδα. Τέλος, η πρόοδος ως προς ε, την προσθήκη του περιβάλλοντος ε, και ε, του η δράση για το κλίμα δεν είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό το βλέπουμε στην πρόσφατη έκθεση του Ελεκτρικού Συνεδρίου για το πρασίνισμα και οι οικονομικέ διαφορέ ανάμεσα στι περιοχέ Υπέθρου και άλλε περιοχέ έχουν επίση μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν. για τα απορίσματα και τα κριτήριά μας για την κοινή γεωργική πολιτική. Πρώτον, Αυτό την προσοχή σας στην προσέγγιση που υιοθετήσαμε. Ξαναλέω, δεν είμαστε εμείς πολιτικό σώμα και άρα θα πρέπει να βασιστούμε σε τεχνικά κριτήρια, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ένα έγγραφο, μια πολιτική, ένα πρόγραμμα κτλ. Και το μοντέλο που χρησιμοποιούμε εν είναι το εξή και ε, ε, ταχύτατα θα σας το εξηγήσω. Έτσι εμείς αναλύουμε τις ανακοινώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτον, πρέπει να προσδιοριστούν οι ανάγκες που εξυπηρετεί μια δημόσια πολιτική. Κατόπιν, οι ανάγκες αυτές θα, ε, από αυτές τις ανάγκες απορρέουν και στόχοι. Και για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους ε, παρέχουμε μια συγκεκριμένη προσπάθεια input και συγκεκριμένες διαδικασίες με τα input ε, ε, και, την, ε, και τις διαδικασίες καταλήγουμε στα output, στα παραγόμενα αποτελέσματα, εξετάζοντας και τους εξωτερικούς παράγοντες. Αυτό είναι το μοντέλο που χρησιμοποιούμε εμείς. Έτσι αναλύσαμε και την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε σχέση με στόχους και ανάγκες. Υπάρχουν ε, οι απαιτούμενες προφορές για να προσδιορίσουμε ειδικέ ανάγκες και να δικαιολογήσουμε τωρινές δαπάνες κυνηγής γεωργικής πολιτικής. Όμως, κατά τη γνώμη μας, δεν υπαρκούν οι πληροφορίες. Δεύτερον, η έννοια της ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας προϋποθέτει ε, μεγαλύτερη σαφήνεια. Για μας δεν έχει διευκρινιστεί το ζήτημα, οπότε η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να ανταποκρίνεται στις μακροπρόθεσμες τάσεις. Ποιες, ποιοι είναι οι στόχοι. Αυτοί οι στόχοι τη κοινή γεωργική πολιτική δεν είναι παρκώς σαφείς και συγκεκριμένοι. Στο την προσοχή σα. Οι δαπάνε ε, στον τομέα αυτό στο παρελθόν και σας υπενθυμίζουμε ότι λαμβάνουμε υπόψη την τρέχουσα ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα στοιχεία της. Λοιπόν, αυτή η ανάγκη που εντοπίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια σε σχέση με άλλους στόχου, στα πλαίσια άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα inputs, ε, την κατανομή των χρηματοδοτικών ε, ταμείων δεν βασίζονται σε επαρκή αξιολόγηση της ε, ε, βασικής ανάγκης ε, παραγωγής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Επίσης, στην νέα κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να έχουμε ταχύτερα με πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες. Χρειάζεται συνέπεια ανάμεσα στην κοινή γεωργική πολιτική και άλλες πολιτικές και ανάμεσα στα επιμέρους όργανα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα πρέπει να απλουστεύουμε, αλλά όχι εις βάρος αποτελεσματικότητας. Τέλος. Ως προς τις διαδικασίες. Η εκπόνηση ε, της μελλοντικής ε, γεωργικής πολιτικής ε, είναι χρονοβόρα διαδικασία. Το υπενθυμίζω. Και Έχουμε ανησυχίε σε σχέση και με την παραγόμενη αξία και του εξωτερικού ε, κινδύνου. Δηλαδή, οι τωρινοί δείκτε δεν επαρκούν για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των ενών πολιτικών. Χρειαζόμαστε σαφή σύνδεση ανάμεσα ε, στην αξιολόγηση αντικτύπου και στην επίτευξη των στόχων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ε, σύνδεση ανάμεσα στα χρήματα που ξοδεύουμε και την επίτευξη των προσδιορισμένων στόχων. Και σε δηλώσει που έχουμε κάνει στο παρελθόν, ξεκαθαρίζουμε ότι πρέπει να προσδιορίσουμε ποιοι είναι οι υπόλογοι, πώ απαιτείται η ευθύνε στην κοινή γεωργική πολιτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπενθυμίζουμε στου νομοθέτε μέσα σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο για το μέλλον τη κοινή γεωργικής πολιτική ότι αυτό είναι βασικό ζήτημα. Αλλά όπω είπα ήδη πολλέ φορέ δεν είναι πολιτικό όργανο το ελεγκτικό συνέδριο και άρα δεν μπορεί να καταθέσει συγκεκριμένε προτάσει για το μέλλον. Πλην όμως θεωρούμε πως το ελεγκτικό συνέδριο έχει την ευθύνη να εισηγηθεί συγκεκριμένα κριτήρια στους νομοθέτες για να μπορούν να αξιολογούν αν οι μελλοντικέ προθέσει είναι ικανοποιητικέ, επαρκούν και αν πρέπει να εφαρμοστούν ναι ή όχι. Τα κριτήρια περιστρέφονται γύρω από κάποιες βασικές ιδέες που σας περιέγραψα. Ξανά, οι ανάγκες. Στην νέα γεωργική πολιτική θα πρέπει να ζητούμε σε συγκεκριμένα τεκμήρια για να εντοπίσουμε τις ανάγκες μας. Η προσθέμενη αξία θα ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να αποδεικνύεται. Οι προτάσεις κοινή γεωργική πολιτικής λαμβάνουν υπόψη μακροπρόθεσμες τάσεις, είναι σαφείς σε σχέση με την κατανομή των, του αντικτύπου και ανταποκρίνονται αυτά για τις ανάγκες. Σε σχέση με τους στόχους, οι στόχοι προσδιορίζονται με σαφήνεια και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στην ε, μακροπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο όραμα για την ε, κοινή γεωργική πολιτική. Μεταφράζονται σε μετρήσιμους στόχους ως προς ε, τον αντίκτυπο και το αποτέλεσμα, συνάδουν με την, ε, τις συνολικούς και επιμέρους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τομεακούς στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις. Τα κονδύλια κατανείμονται βάσει της αξιολόγησης των αναγκών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων ε, οι δαπάνε είναι στου τομεί όπου μπορούμε να αναμένουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Εφαρμόζονται οι πολιτικές με όργανα που είναι τα αποτελεσματικά και βασιζόμαστε σε συγκεκριμένα τεκμήρια. Υπάρχει συνέπεια ανάμεσα στην κοινή γεωργική πολιτική και άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκή Ένωση και στα, ανάμεσα στα επιμέρου όργανα τη κοινή γεωργική πολιτική, Οι εφαρμοστικοί κανόνε είναι απλοί και δεν ε, θέτουν ε, εν κινδύνο την αποτελεσματικότητα σε σχέση με το κόστος των μέτρων. Έχουν γίνει ρυθμίσεις για τη μετάβαση ε, στο νέο μοντέλο χορήγησης της στήριξης και σε σχέση με την παραγόμενη αξία και τους εξωτερικούς παράγοντες ένα νέο σύστημα συνδέει τους στόχους και τον αναμενόμενο αντίκτυπο. Υπάρχει σαφή σχέση ανάμεσα στα χρήματα που εκμεταμιεύονται από τον προπολογισμό και την των ε, εκ των προτέρων προσδιορισμένων στόχων ε, παρακολουθούμε τους εξωτερικούς ε, παράγοντες και προσαρμόζουμε αναλόγως την πολιτική όπου δει και τέλος σε σχέση με την απόδοση ευθυνών στις νέες προτάσεις για την κοινή γεωργική πολιτική ε, ε, είναι ενισχυμένο αυτό το σύστημα σε σχέση με την απόδοση ευθυνών και την αλυσίδα ελέγχων. Αυτά είναι κριτήρια για την αξιολόγηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Και στο ενημερωτικό δελτίο μπορείτε να δείτε πώς... Ε, αναλύουμε τους λόγους και τη βάση για που εξηγούν για ποιο λόγο εμείς εισηγούμαστε αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια για την ε, αποτίμηση των προτάσεων για την μελλοντική γεωργική πολιτική. Τώρα, ε, ο ρόλος ε, των συνομοθετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να ε, διορθώσουν, να αναθεωρήσουν, να προσαρμόσουν αυτά τα κριτήρια. Όμως λέω, κατά πάσα πιθανότητα, όταν το Μάιο-Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει τις προτάσεις της, εμείς τέτοιου είδους κριτήρια θα χρησιμοποιήσουμε για να αξιολογήσουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο συγητής μας είναι ο κ. Τσέλερ. Κύριε Φιγερέιδε, επιτρέψατε μου να σας πω το εξής. Ε, ε, σήμερα λάβαμε το έγγραφο στις 3 και 22 ε, δεν υπήρξε καμία δυνατότητα συνεπώς να το διαβάσουμε και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε τα κείμενα νωρίτερα εφόσον κάνουμε συζητήσεις πραγματικά βαρύνουσα σημασίας. Ο κύριος Τσέλερ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και ακούω τις κραυγές των συναδέλφων από την Επιτροπή Γεωργίας αλλά και από τις χώρες μέλη. Τι ανακατεύεται τώρα το ελεκτικό συνέδριο στα περιεχόμενα της συνέχισης της κοινής, αγροτικής, ε, κοινής γεωργικής πολιτικής. Παρ' όλα αυτά είμαι εξαιρετικά ευγνώμων προς τον, συνάδελφο κύριο, προς τον κύριο Φιερέδο και προς τους συναδέλφους του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υποβολή αυτού του γράφου. Γιατί ε, οι έλεγχοι που έκαναν ε, μας έδωσαν μία εποπτεία όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της ε, κοινή ε, γεωργικής πολιτικής. Και βεβαίως μας επιτρέπουν να καταλήξουμε σε μία αξιολόγηση της ΚΑΠΑ μέχρι τώρα, ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε προτάσεις για τη μελλοντική της διαφόρφωση. Ο κόσμος περιστρέφεται, τα πράγματα αλλάζουν και η Επιτροπή θα πρέπει να δει πού θέτει την ε, έμφαση των ε, προτεραιοτήτων της. Οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Γεωργίας ε, θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν και πώς θα επιμεριστούν τα μελλοντικά κονδύλια. Η Γεωργία καταλαμβάνει 40% του ευρωπαϊκού προπολογισμού και θα πρέπει να δει το ερώτημα κατά πόσο όλα αυτά πραγματικά είχαν νόημα. Και θα ήθελα να τονίσω δύο φράσεις από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ή από το κατάλογο των θεμάτων όπου αναφέρεται ότι τα κονδύλια της ΚΑΠ επιμερίζονται στις χώρες μέλη υπό τη μορφή εθνικών χαρτοφυλακίων τα οποία δεν ορίζονται στη βάση των αναγκών των χωρών μελών ούτε, δεσμεύσεις, ούτε δεσμεύσεις για συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ε, η μέθοδος αυτή εγκαιμονεί κάποια ρίσκα όσον αφορά τις μελλοντικέ δαπάνες και διαπιστώνουμε ότι ε, δεν υπάρχουν επαρκείς αιτιολογήσεις όσον αφορά τον, την κατανομή των κονδυλίων, ε, τα οποία θα πρέπει να επιμερίζονται εκεί όπου ε, δαπανώνται σωστά και ο ΣΑ ορίζει ε, ένα performance budgeting, ένα προπολογισμό ο οποίος ε, επιμερίζει τα χρήματα ε, βάσει των αποτελεσμάτων. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συμπελάβουμε αυτές τις σκέψεις στη δική μας συζήτηση και να δούμε ότι στο πλαίσιο μιας ε, γεργίας η οποία αλλάζει, στο πλαίσιο μιας εκβιομηχάνησης και όπου υπάρχουν όλο και μεγαλύτερες εκτάσεις που γίνονται αντικείμενο κερδοσκοπίας ε, και υπάρχει και μια διεύρυνση των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παράγονται και κάποια προϊόντα τα οποία ε, σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας, ενέργειας. Και νομίζω ότι ήταν ε, σωστή και η παρατήρηση του ελεγκτικού συνεδρίου ότι είμαστε καθαροί εξαγωγής σε σχέση με τις εισαγωγές μας. Και αν δούμε τι γίνεται στην γεωργία μας, σε αντίθεση με τη γεωργία σε αναπτυσσόμενες χώρες, Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ελλείμματα τα οποία θα πρέπει να διορθώσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για το κείμενό σας. Η Επιτροπή ήδη στην ε, παρούσα περίοδο προσπάθησε να στρέψει τα πράγματα προς την ορθή κατεύθυνση και ήταν ε, αυτοί που συναποφάσισαν στην ε, δικασία της νομοθεσίας, οι οποίοι ε, πέσυραν κάποια σημεία εδώ, αλλά νομίζω ότι η συζήτηση αυτή θα πρέπει να συνεχίσει. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Τσέλερ, κυρία Πρόεδρε, ε, μέλη ε, αυτή τη Επιτροπή, ε, κύριε Φιγερέιρο, αγαπητοί συνάδελφοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Χαιρετίζουμε αυτό το κείμενο γιατί πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και αξιόλογο input στη συζήτηση, στη συζήτηση και έχει σαν στόχο ε, τελικά την αποκριστάλλωση σε κάποιες νομοθετικές ε, προτάσεις ε, το Μάιο αυτού του έτους. Κάθε συμβουλή και κάθε εισφορά στη συζήτηση αυτή θεωρώ ότι μπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμη. Είμαστε ευτυχείς που διαπιστώνουμε ότι το συνέδριο στο κείμενό του αναγνωρίζει ότι η ανακοίνωση ανταποκρίνεται σε πολλέ ε, συστάσεις που έγιναν σε παλιότερε εκθέσει του ελεγκτικού συνεδρίου. βεβαίω, όχι, ε, δεν ανταποκρίνεται σε όλε, αλλά σε αρκετέ από αυτέ. Και αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει μια ευαισθησία εκ μέρου της επιτροπή όσον αφορά τι προτάσει αυτές. Όπως είπε ο κύριος ε, Τσέλερ, τελικά θα είναι οι συνομοθέτες αυτοί οι οποίοι θα χαράξουν την πολιτική όπως έχει γίνει στο παρελθόν δεν υπάρχει καμία, και όπως έχει υποθεί δεν υπάρχει καμία πρόταση της Επιτροπής στην οποία το Κοινοβούλιο να έχει αφήσει άθικτη ούτως ώστε να φύγει έτσι όπως ήρθε. Η ανακοίνωση προσπαθεί να εισαγάγει ε, κάτι το οποίο αναφέρθηκε κατά επανάληψη στη συζήτηση αλλά και στην προηγούμενη συζήτηση για το προηγούμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης προσπαθεί να πετύχει μια νέα ισορροπία ε, ορίζοντας εκ νέου το ρόλο των ε, διαφόρων των δρόντων στην διαδικασία αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες ε, μέλη και η εισαγωγή ενό νέου μοντέλου, το οποίο δεν θα πρέπει να θεωρείται απλώς και μόνο σαν ένα εργαλείο να δοθούν όλες οι εξουσίες στις χώρες μέλη, αλλά σαν εργαλείο επαναπροσανατολισμού των πολιτικών προς στόχους που απομακρύνονται από τον αποκλειστικό προσανατολισμό προς ε, κανόνες, ε, διαδάξεις και διαδικασίες που ίσχυαν στο παρελθόν. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Ε, δηλαδή δεν θα συζητούμε ε, Πρωτήσω κατά πόσο κάποια μέτρα ήταν ορθά και κατά πόσο υπήρξε εφαρμογή συμμόρφωση με ορισμένου κανόνε, αλλά θα συζητούμε αυτής εξ αρχή ε, ποιοι είναι οι στόχοι που θέλουμε να ακολουθήσουμε ε, και κατά πόσο θέλουμε να κινηθούμε προ αυτή την κατεύθυνση. Και σε ποιο μέτρο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Λοιπόν, αυτό ε, προϋποθέτει ότι θα προσδιορίσουμε εκ νέου τους στόχους γιατί είναι ε, πολύ διαφορετική κατάσταση στις επιμέρους περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα η κατάσταση της Γεωργίας και άρα θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν ένα ενισχυμένο ρόλο για να δουν επιτόπου ποιες είναι οι ανάγκες και να ορίσουν τους στόχους τους αναλόγους. Η Επιτροπή επομένως θα ελέγξει το κατά πόσον ορθά έχουν τεθεί οι στόχοι από πλευρά κρατών μελών σε διάλογο μαζί τους. Άρα μαζί θα προγραμματιστούμε για την καινούργια ΚΑΠ και θα δούμε επί τόπου τι ισχύει σε σχέση με το πρόγραμμα και κατά πόσον οι στόχοι επιτεύχθηκαν. Άρα και οι στόχοι και η μέτρηση των επιδόσεων θα γίνουν στους επιδοκρατών μελών η σχέση με τους δικαιούχους θα απλουστευτεί, κάνουμε ό,τι μπορούμε, να προσθέσουμε την ε, πολιτική, να μην έχουμε πολυνομία όπως σήμερα. Και θα απόκειται στα κράτη-μέλη να θεσπίσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο στα πλαίσια δηλαδή της δικής του ένωμης τάξης και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουμε και την σύγχρονη τεχνολογία για να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή των γεωργών. Η σημερινή δομή της διακυβέρνησης της ΚΑΠ θα πρέπει να συνεχίζει να ισχύει μια και δουλεύει έβρεθμα και μιλούμε για τους οργανισμούς πληρωμής, για τις άλλες συναρμόδιες αρχές, όλα αυτά συνεχίσουν Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη και όταν κάνουμε και τον οικονομικό έλεγχο όσον αφορά τους, τους οργανισμούς πιστοποίησης που θα έχουν ακόμα πιο αναβαθμισμένο ρόλο. Άρα, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να γίνει μια στροφή όσον αφορά τις αρμοδιότητες και να υπάρχει ένα αυθεντικά κοινό πλαίσιο, να είναι ξεκάθαρο και να μπορούμε να κυνηγήσουμε πάνω από έναν στόχο την αποτελεσματικότητα της ε, πολιτικής, την απλούστευση, όλους μας στόχους ταυτόχρονα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι θετικά όσα λέει το ελληνικό συνέδριο που λέει με τη σειρά του ότι θέλει να κινηθεί προς τη δική μας πρόταση και λέει παραπέρα ότι αν εφαρμοστούν αυτά όπως πρέπει το θα είναι πιο αποτελεσματική η κοινή αγροτική πολιτική που αυτό και εμείς θέλουμε να πετύχουμε. Όσον αφορά το ενημερωτικό σημείο μας λέει ε, πώς θα πετύχουμε ε, από πλευράς ε, ε, επιστημονικής ε, τεκμηρίωσης, βιωσιμότητας, ε, νέους στόχους, λέει για στεγανούς ελέγχους, αξιολογήσεις, ε, να, ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο διαδικασία απόδοσης ευθυνών, Δηλαδή όλα αυτά καταλήγουμε στο ότι είναι σημαντικά. Θα πρέπει να συντρέχουν, άλλο το νέο σύστημα δεν θα πετύχει αυτά που οφείλει. Δύο λόγια τώρα όσον αφορά μια προβληματική που ξεκίνησε και για το προηγούμενο θέμα, δηλαδή για τα βασικά στοιχεία, τα key data και τι γίνεται σε σχέση με το εισόδημα των γεωργών. Εκεί πολλές φορές έχουμε έντονες συζητήσεις και με το ελληνικό συνέδριο θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο εισόδημα των γεωργών και όχι των οικοκυριών. Πρώτα-πρώτα γιατί ο στόχος της ε, συνθήκης είναι η γεωργική δραστηριότητα. Και, και διότι η συνθήκη θεωρεί τη γεωργική πολιτική είναι οικονομική πολιτική και όχι κάποια κοινωνική πολιτική. Ε, αυτό το πράγμα θεωρείται η γεωρική πολιτική παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε όλοι αυτοί οι στόχοι έχουν σχέση άμεσα με την παραγωγικότητα, την, τον εξορθολογισμό κλπ. για την γεωργική παραγωγή. Τώρα όσον αφορά την υποστήριξη του 92 για προϊόντα και παραγωγούς θέλουμε να είναι πιο πολύ προσανατολισμένοι στην αγορά, να έχουμε το Δικτύο Ασφαλείας του Εισοδήματος και εδώ επομένω να εστιαζόμαστε στην εκμετάλλευση και όχι στο νοικοκυριό. Και τέλος, και κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτό δεν ισχύει, δεν έχουμε αρκετά δεδομένα εισοδήματος, μόνο πέντε κράτη-μέλη μας στέλνουν στοιχεία για το εισόδημα. Είναι πολλοί παράγοντε που επηρεάζουν το εισόδημα πέραν τη γεωργία. Οπότε και αυτά είναι αρμοδιότητα εθνική. Φορολογία, νομοθεσία, ε, συντάξεις και άλλα. Όλα αυτά είναι εθνικές αρμοδιότητες, άρα δεν μπορούμε να ανακατευτούμε σε αυτά. Δεν κατακλείδη. Σωστά τα είπε το κύριε ότι οι δαπάνε είναι σταθερές της κάπου πολλά χρόνια. Σωστό. Με τις τρέχουσες τιμές. Αν όμως δείτε σε σταθερές τιμές τις δαπάνε, δηλαδή με την ΆΤΑ, τότε βλέπετε ότι έχουν μειωθεί οι δαπάνε στη σχετική περίοδο. Και θα μειωθούν ακόμα περισσότερο κατά την επόμενη περίοδο. Άρα δεν ισχύει το ότι όλο ένα και πιο ακριβή καθίσταται η ΚΑΠ από πλευράς του πόσο πρέπει να δαπανά. Μάλλον μειώνει τη δαπάνη παρά αυξάνεται. Ευχαριστώ. Ε, δεν ξέρω για ποια άλλε ε, παραγωγέ εισοδήματο μιλάμε. Έχω την εντύπωση ότι μόνο με αυτό ασχολούμαστε ακόμη για τα είδη φούρνου. Ε, παρακαλώ. Κύριε Χόλμπουχ. Ε, κύριε Τσέλερ, είπατε ότι το 20% το, 40% ε, του προϋπολογισμού εξακολουθεί να διοχετεύεται στη Γεωργία. Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτά είναι για τον ενωσιακό προϋπολογισμό, είναι πολύ χαμηλότερα τα εθνικά κονδύλια. Ε, και κάνουμε ένα top-up στη Γεωργία, παραδείγματο χάρη, είναι με μικρή υποστήριξη μέσα από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και ο βασικός προϋπολογισμός είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όταν μιλάτε για φόρους εξαγωγής και ότι αυξήθηκαν ε, τα εισοδήματα. Τι λαμβάνουν από αυτό οι γεωργοί. Για τα μεταποιημένα προϊόντα είμαστε καθαροί εξαγωγής ε, και για τα, τους εισαγωγείς είναι για τις πρώτες ύλες, μη μεταποιημένα προϊόντα, αν κατάλαβα καλά. Μόνο ένα παράδειγμα για να καταλάβετε για το πράγμα μιλάω. Κατά την κρίση γάλακτος ε, εξήγαμε ε, πολύ περισσότερη σκόνη γάλακτος ε, και χάσαμε με, πολλά ε, εισοδήματα από το, το ίδιο το γάλα, δηλαδή 3,2 δισεκατομμύρια τόνους που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Καταλαβαίνετε ότι οι γεωργοί τι παίρνουν από αυτά, δεν τα πηγαίνουν στη, στη, στον Παναμά και στα νησιά Κέιμαν, επιστρέφουν αυτά τα χρήματα στην ε, τοπική γεωργία, στην οικονομία. Οπότε θα πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Είναι πολλά τα προβλήματα, πολλέ οι προκλήσεις, πρέπει να προστατεύσουμε το κλίμα, την, ε, ε, το ευσύν των ζώων, ε, να μειώσουμε τα ε, ζυζανιοκτώνα. Όλα αυτά κοστίζουν χρήματα και θα πρέπει να είναι βιώσιμες προτάσεις μας για την ε, γεωργία λοιπόν γιατί πράγμα χρηματοδοτούμε και ποιος τελικά παίρνει αυτά τα κονδύλια. Αυτά είναι βασικά ερωτήματα και πρέπει να τα απαντήσουμε. Ναι, ναι, συμφωνούμε. Οι μεγάλοι και οι πλούσιοι, αυτοί που επενδύουν σε μεγάλες γεωρικές εκμεταλλεύσεις, γιατί ξέρω το μάνα εξ ουρανού έρχεται από την Ευρώπη, δεν πρέπει να συνεχίζουν να υποφελούνται ε, και ε, δεν θα πρέπει ε, να γίνεται αυτό εις βάρος των μικρών παραγωγών και να προσπαθούν να εμποδίζουν κάθε μεταρρύθμιση που είναι εις βάρος τους. Θα θέλω να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Φιγκρέη, τον ακούσουμε σύντομα και τον εισηγητή και ο ε, εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσω θα μπορούσε να μα δώσει ε, κάποιε απαντήσει. Μπορείτε να μα στείλετε και γραπτό ακόμη καλύτερα. Δηλαδή, από τι εξαγωγέ, ε, πόσα πηγαίνουν στι αναπτυσσόμενε χώρε, ποιο ποσοστό, διότι χτε. κάναμε μια δύσκολη συζήτηση για γιατί η, κατάσταση είναι όπως είναι και αν δεν είχαμε τη συγκεκριμένα δεδομένα θα είχαμε κάνει και εμείς το ίδιο λάθος σε σχέση με την αναπτυξιακή πολιτική. Εγώ στις Ευρωπαίκες Επιτροπές. Δύο σύντομα σημεία θέλω να μας απασχολήσουν. Πάρα πολύ λίγες εξαρτημένες από τις τις χώρες. Όμως εισάγουμε περισσότερα από τις χώρες παρά από ΙΠΑ, Καναδά, Κίνα και Ιαπωνία μαζί. Άρα είμαστε πηγή εισαγωγών για τις χώρες αυτές, αλλά λίγα πάνε εκεί. Λίγα προϊόντα. Σας δώσω στοιχεία, σας στείλω στοιχεία. Τώρα στην ανακοίνωση, κοιτάξτε, θα βρείτε τα σχετικά στοιχεία και το ότι 72% της στήριξης πάει σε ε, μεταξύ 5 και 250 εκταρίων. Οικογενειακές δηλαδή εκμεταλλεύσεις. Τίποτα το περίεργο. Υπάρχουν βέβαια κάποιες μεγάλες εκμεταλλεύσεις που παίρνουν ε, στήριξη μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις Έχουμε, ας πούμε, 10.000 εκταρίων επιχειρήσεις που μπορεί να είναι επικερδείς, αλλά έχουμε πάρα πολλές μικτής εκμετάλλευσης, δηλαδή και με γεωργικά προϊόντα και με κτηνοτροφικά. Άλλα έχουν σχέση με συνεταιρισμούς, άλλες ε, εκμεταλλεύσεις και οι ίδιοι οι γεωργοί, οι δουλεύουν εκεί. Επομένως, συνήθως τα, πράγματα ε, χρειάζονται μεγαλύτερη ποικίλια από ότι αυτό το 80-20, το κλασικό που λέγεται. Και αυτό θα πρέπει να προβληθεί. Πρόεδρος. Ειλικρινά θα ήθελα να το αφισβητήσω γιατί διαπιστώνουμε ότι 90% των εισοδημάτων πηγαίνουν στο 10% των γεωργών. Εάν δούμε λοιπόν τι γίνεται ε, και μπορούμε να το κάνουμε τους αριθμούς της Επιτροπής, ε, δεν καταλήγουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Και βεβαίως είμαστε διατεθειμένοι να παρακολουθήσουμε κάθε παρουσίασή σας με PowerPoint και βεβαίως θα θέλαμε να καλέσουμε και το ελεκτικό συνέδριο. Γιατί το ερώτημα ποιος παίρνει τα χρήματα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε αυτή την ερώτηση. Ε, τώρα έχουμε έρθει σε... βρισκόμαστε σε χρονική πίεση. Δύο συνάδελφοι να πάρουν το λόγο παρακαλώ να είστε σύντομοι. Γιατί στις 5.30 πρέπει να αρχίσει η συνεδρία των συντονιστών. Ο συνάδελφος κ. Φλένιγκερ. Όλα εξαρτώνται από το πώς ε, γίνονται οι στατιστικές. Γιατί όταν λέτε ότι η στήριξη των εισοδημάτων πηγαίνει στους μικρούς ε, καλλιεργητές, ε, για παράδειγμα 250 εκτάρια. Ε, στη δική μας χώρα ε, θα παίρναμε ε, λιγότερα χρήματα από ότι κάποιος ο οποίος έχει πέντε εκτάρια. Ε, το θέμα είναι η κατάσταση ποικίλει από χώρα σε χώρα. Ε, βεβαίως πηγαίνουν πάρα πολλά χρήματα στους πλούσιους καλλιεργητές. Και στο τέλος αυτής της ε, θητείας εγώ είμαι σίγουρος ότι θα αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα γιατί τα κατεστημένα συμφέροντα θα κατησχίσουν, θα υπερσχίσουν και πάλι και τα χρήματα θα μείνουν στις ίδιες τσέπες. Η κυρία Νόχερ εάν μιλάμε για μια στήριξη εισοδημάτων στον πρώτο πυλώνα και αυτός ο ορισμός στήριξη εισοδήματος δεν είναι δική μου επινόηση τότε πρόκειται για μια κοινωνική μεταφορά κονδυλίων. Και αν πρόκειται για μια κοινωνική μεταφορά κονδυλίων, θα πρέπει να συναρτάται από τις ανάγκες των ατόμων. Γιατί δεν υπάρχουν κοινωνικέ μεταφορές ανεξάρτητα από τι ανάγκε των ατόμων. Και επίσης θα πρέπει να συναρτάται με το πόσοι άνθρωποι χρήζουν αυτής της ε, ενίσχυσης ε, και ε, μια ακάλυπτη κοινωνική μεταφορά υπάρχει μόνο στον πρώτο πυλώνα και θα πρέπει κατεπηγόντως να καλυφθεί. Λοιπόν, πρόεδρε, θα το λάβω υπόψη μου. Βλέπω ότι όλοι χαίρονται για την συνέχιση της συνεδρίασης αύριο. Ο κύριος Φεγγερέιδο έχει και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, Θέλω να σας πω ότι τολμηρά να σας πω τα εξής και σύντομα. Πρώτα πρώτα. Μεγάλη μου ικανοποίηση βλέπω ότι θεωρεί θετικέ τι τάσει μα η Ευρωπαϊκή Τροπή. Αυτό είναι συμβολή μα στην προβληματική. Αν δηλαδή το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι χρήσιμο το έγγραφο, αυτό θα μας ικανοποιήσει πάρα πολύ. Και έτσι όπως πάει το πράγμα, εάν το Κοινοβούλιο θέλει ενεργότερο ρόλο για το ελληνικό συνέδριο, εμείς είμαστε στη διάθεσή σας. Απλώς ζητήστε το. Τώρα. Εγώ θέλω το εξή να κρατήσουμε από αυτή τη συζήτηση. Πολλά θα μπορούσε να πει κανεί, αλλά εδώ και τώρα σας τονίζω ως εξωτερικός ελεγκτής ότι να σταθούμε στο εξής. Συμφωνώ 100% με αυτή την στροφή. προς το να έχουμε ως επίγειδος προσοχής μας τις επιδόσεις και την αξιολόγηση των επιδόσεων ως ε, οικονομικός ελεγκτής, ως μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Πρέπει να απευθυνθώ στον νομοθέτη να λάβει υπόψη το θέμα της συμμόρφωσης γιατί αυτά τα πράγματα πάνε χέρι-χέρι η επίδοση και η απόδοση σε σχέση με την συμμόρφωση αφού πέρασε η εποχή που προσέχαμε μόνο την συμμόρφωση τώρα δεν είναι δυνατόν να την αγνοήσουμε ολοσχερός. πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα αφορά τι ε, υπηρεσίε μα που γίνουν την πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Άρα και επιδόσει και συμμόρφωση. Ε, ευχαριστούμε. Ναι, ρίξα το μπαλάκι τώρα σε εμά. Ε, άρχισε το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, ε, είμαστε Δηλαδή δεν μπορούμε με τίτλους ε, να ε, βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα. Όταν ε, μιλάμε για τους εξαγωγείς, ναι, μιλάμε για τη βιομηχανία και όχι για τους, ε, μικ, τις μικρές εκμεταλλεύσεις ε, και οι ιδιοκτήτες αυτών των μεγάλων ιωρικών εκμεταλλεύσεων δεν είναι εκεί γιατί καταλαβαίνετε ότι πηγαίνουν στις πόλεις. Δεν είναι καν στην Ήπεθρο γιατί στις πόλεις είναι η βιομηχανική ανάπτυξη. Οπότε δεν μιλάμε για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, στην Ήπεθρο και δεν είναι ότι εργάζονται για μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Όχι, μιλάμε για βιομηχανίες που βρίσκονται στις πόλεις. Εμίλ, μας ε, είπατε για την περίπτωση του γάλακτος. Ε, λοιπόν, ε, είχαμε την, ε, το συλλαλητήριο ε, των γυναικών των γαλακτοπαραγωγών και στην Ιρλανδία οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας μας είπαν «Μα επιτέλους να θέλουμε να ξεφορτωθούμε τις ποσοστώσεις γάλακτος, απελευθερώστε μας γιατί θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό μας, θέλουμε να παράξουμε περισσότερα για να έχουμε και περισσότερα κέρδη, να έχουμε αυτή τη δυνατότητα». Καταλαβαίνετε, υπάρχει μια διαφοροποίηση και γι' αυτό, όπως είπε η κυρία Μίγλε θα πρέπει κατά περίπτωση ε, να εξετάσουμε τη, την κατάσταση και ε, ε, με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να διαμορφώσουμε τις συζητήσεις μας. Ε, πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ε, φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίας, στο τέλος της ανοιχτής συνεδρίας. Σας ευχαριστώ για ε, τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή σας. Ε, κυρίσω τη λήξη της ε, δημόσιας συνεδρίας για να αρχίσουμε τη συνεδρία των συντονιστών. Ευχαριστώ. Αύριο στις αρχίζουμε με τις ψηφοφορίες για τις εξωτερικούς οργανισμούς, ε, τις κοινέ επιχειρήσεις ε, και τους λοιπούς οργανισμούς. Ευχαριστώ.